έναρξη της συνεδρίασης. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κοέλιο με θέμα δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Κοέλιο για τέσσερα λεπτά. Obrigado, Sr. Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπη Μπιενκόφσκα, συνάδελφοι. Εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειε και περιμένουμε να δούμε πώς προχωράει η υλοποίηση από τα κράτη-μέλη. Αξιολογούμε λοιπόν αν πήγε καλά ή όχι και αν ακολουθήθηκαν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Να θυμίσουμε ότι οι δημόσιες προμήθειες είναι πολύ σημαντικές για την εσωτερική αγορά. Ε, υπάρχει και το σχετικό στρατηγικό πλαίσιο για να προωθηθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και η καινοτομία. Οι δημόσιες συμβάσεις ε, αποτελούν σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία μας, πάνω από 12 δις ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι 280.000 δημόσιες αρχές ε, παράγουν το 14% και χειρίζονται το 14% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με έργα, υποδομές και δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει ε, να προσφέρουμε δημόσιε υπηρεσίε υψηλή ποιότητα και όλα αυτά βεβαίω εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία δημόσιων προμηθειών που θα εγκρίνουμε, προκειμένου να είναι αποτελεσματική και διαφανή. Η έκθεσή μα λοιπόν προσπαθεί αυτή την ανάγκη ακριβώ να υπογραμμίσει. Η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να, είναι να προτείνει ένα πακέτο μέτρων μη νομοθετικών, όπω έχει γίνει ήδη με δύο ανακοινώσει και ε, μία δήλωση για τη διαδικασία των δημόσιων προμηθειών. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερου νόμου, αλλά καλή εφαρμογή των κανόνων που ήδη ε, διαθέτουμε Γι' αυτό, ε, ολοκληρώ, γι αυτό εγκρίναμε ένα σύνολο από που ενέκρινε η Επιτροπή τη Εσωτερική Αγορά. Οι οδηγίε που εγκρίθηκαν το 2014, συνάδελφοι, δεν είναι απλώ ένα εργαλείο για να ε, εγκρίνουμε την ε, διαδικασία δημόσιων προμηθειών για έργα, αγαθά και υποδομέ. Είναι και για έργα καινοτομία, τη ε, οικολογική και κυκλική οικονομία και τη συμμετοχική βιώσιμη ανάπτυξη. Βεβαίω, είναι απογοητευτικό ο ρυθμό από τον οποίο τα κράτη-μέλη μεταφέρουν την οδηγία και πολλέ φορές ε, έχουν ε, αντιμετωπίσει και διαδικασία επιπαραβάση. Θα πρέπει λοιπόν να πάψει ο προστατευτισμός και να μπορέσουν εύκολα να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περισσότερη απλούστευση και περισσότερη διαφάνεια. Ε, δεν θα πρέπει απλώ να είναι μειοδοτική διαγωνισμή και να επιλέγεται όποιο προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε μια σειρά από μέτρα που μπορούν να υλοποιηθούν και δικαιολογούνται για να έχουμε ποιοτικά ε, έργα και υπηρεσίες. Το λέω στην εδάφιο 12 και 13. Ε, επίσης θα πρέπει στην παράγραφο 38 επίσης να προβλέψουμε την ε, σύμβαση, την υποδιέρεση της σύμβασης σε παρτίδες. Επίσης και στις παραγράφους 33 και 41 μιλούμε για τα αξιόπιστα στοιχεία και την πρόσβαση στη δημοσία και μετά για τις παραγράφους 26 ε, και άλλες μιλούμε για την ψηφιοποίηση και για την ε, χρήση και την πρόθεση της καινοτομίας σε παραγράφους 24 και αλλού. Επίσης στην παράγραφο 53 και 57 έχουμε μνήες για την ε, ανάπτυξη πανεπιστημιακών μαθημάτων σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο στο σχετικό θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη δεοντολογία, όπως λένε και οι παράγραφοι 15 και 20, και να ακολουθείται από όλους στη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και του ε, συναδέλφου Χιώδη που συνεργάστηκαν για τη σύνταξη τη έκθεση αυτή, καθώ και του συναδέλφου των Επιτροπών ΕΝΒΙ και ΙΝΤΑ. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια σωστή έκθεση για να έχουμε δημόσιε συμβάσει αποτελεσματικέ, αποδοτικέ, να μπορούν να ανταποκριθούν στι προκλήσει που αντιμετωπίζει όλο το τομέα και να πετύχουμε του στατικού μα στόχου, δηλαδή την καινοτομία, την βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, περιβαλλοντική και κυκλική οικονομία. Ε, ελπίζω με όλου του συναδέλφου να εγκρίνουμε την τελική μορφή τη έκθεση για να λειτουργεί εύρυθμα η εσωτερική αγορά με αύξηση των, ε, της λειτουργίας των επιχειρήσεων και να βεβαιωθούμε ότι ε, οι επιστημονικές μας δυνατότητες θα, προωθηθούν και θα καλλιεργηθούν όλες οι δυνατότητες των πολιτών. Στον ονόματος της Επιτροπής το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Μπιανκόφσκα. Ε, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, εισηγητά, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και ακούσατε τα διάφορα στοιχεία, αλλά πέραν αυτών των στοιχείων πρόκειται για ένα μέσο αποφασιστικής σημασίας για να υλοποιούμε την πολιτική μας. Και οι φορολογούμενοι πολλές φορές βλέπουν να μην πιάνουν τόπο τα λεφτά τους, να μην έχουν τις καλύτερες δυνατές ε, δημόσιες κρατικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και τον ε, Νοέμβριο είπαμε να προωθήσουμε αυτή τη δεσμή διότι θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνει μια στροφή σε αυτή την πολιτική μας, τακτική μας. Μπορεί και για κάτι όλος νέο. Είναι κάποια προαιρετικά μέτρα, κάποιες ε, προτάσεις, κάποιες νέες ε, ιδέες και θα πρέπει βεβαίως να κάποιος να το αγκαλιάσει αυτό το όραμα και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι προτεραιότητες θα τάξουμε, θα πρέπει να βρούμε και κάποια μέτρα εφαρμοστικά. Επίσης αναδεικνύουμε πώς θα βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα, τις διάφορες προκλήσεις για το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα, ε, τις ε, επενδύσεις και τελικά όλα αυτά να οδηγήσουν και σε κοινωνική ένταξη. Υπάρχουν τώρα διάφορα πλεονεκτήματα οικονομικά σε σχέση με το πώς θα έχουμε την καλύτερη σχέση κόστους αποτελέσματος, να πιάσουν το είπαμε τα λεφτά για τους συμπολίτε μας, αλλά βέβαια πάντοτε η επιλογή που γίνεται δεν είναι η πιο φθηνή. Το κοινοτικό δίκαιο δεν απαιτεί να είναι το μόνο κριτήριο στους διαγωνισμούς ο καλύτερος μειοδότης. Και είπαμε επομένω ότι έτσι θα πετύχουν πιο εύκολα τους στόχους μας έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, πρακτικά μέτρα, οπότε προτείνουμε και εμείς δράσεις, αλλά και μέτρα τύπου αρρώγηση Έχουμε έξι προτεραιότητες, τάξη, και επιτρέψτε μου να σας τις αναφέρω σύντομα. Πρώτα-πρώτα, καινοτομία, όσον αφορά τις συμβάσεις, επίσης ε, επαγγελματισμός, δεξιότητες για αυτούς που ασχολούνται και επίσης καλύτερη πρόσβαση για τις ΜΜΕ και γενικότερα τις επιχειρήσεις. Επίσης περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα. Καλύτερη χρήση των δεδομένων, χρήση της τεχνολογίας για απλούστευση και καλύτερη διοργάνωση, περισσότερη συνεργασία των επιμέρους αρμοδίων αρχών. Τον Μαρτιό εγκρίθηκε αυτή η δέσμη μέτρων και τον Φεβρουάριο τα συζητήσαμε στο ΕΚΟΒΙΝ. Αναδείξαμε το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συμβάσεις και από πλευράς δημοσιονομικής. Έτσι και αν έχουμε επαγγελματισμό σε αυτές τις συμβάσεις, τότε έχουμε εξοικονόμηση δαπανών. Η ΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης συμφώνησαν. Ελπίζουμε ότι σήμερα αυτή η διαδρομή θα ολοκληρωθεί. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος και θα εγκριθεί η έκθεση της πρωτοβουλίας η δική σας. Έγινε εξαντλητικά συζήτηση, πολλοί από εσά συνέβαλαν. Ο κύριος ε, Κόλιο κράτησε το τιμόνι του πλοίου και έτσι είχε έτσι κατάληξη αυτή η διαδρομή και η προσέγγιση που επελέγει. Και επίσης έχουμε αφορμή να προβληματιστούμε και για το μέλλον. Υπάρχει ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο και όσο το πλήστον είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος για επιμέρους ζητήματα. Να, ενεργητικά ο ρόλος των ΜΜΕ, όπως προείπαμε. Προσοχή πάντως, να μην είμαστε υπερβολικά απεσιόδοξοι όσον αφορά τα προβλήματα συμμετοχής των ΜΜΕ. Η οδηγία πρόσφατα μεταφέρθηκε στο ιστορικό δίκαιο, οπότε θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι ότου η απλούστευση ολοκληρωθεί. Πρόσφατα κάναμε κάποια μελέτη να άρουμε τους τελευταίους φραγμούς όσον αφορά τη συμμετοχή των ε Δεύτερον, τα κριτήρια ποιότητας, στρατηγικές συμβάσεις προμήθειας, μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Άρα υπάρχει έδαφος ε, βελτίωση κατάστασης. Να μην είναι υποχρεωτικό επομένως το θέμα ε, της ε, ελάχιστη ε, τιμής. Πολύ σημαντικό το θέμα της δέσμευσης και η υπερβολοντική πτυχή για αυτές τις συμβάσεις. Άρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι καλύτερες πρακτικές από τις αρμόδιες αρχές. Η ψηφιοποίηση προδεινοφελήσει πάρα πολύ και αυτό το θέμα. Επίσης και η επαγγελματική αντιμετώπιση αυτών των κρατικών δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με όσα είπατε και κάναμε ένα συμπίλημα αυτών των ε, καλύτερων πρακτικών στα διάφορα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να επισημάνουμε σε αυτό το με τα καλύτερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, ε, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πράγματι, οι δημόσιες ε, συμβάσεις αναφέρονται μόνο παρόδο αλλά αυτό είναι λάθος. Σήμερα για τον ανταγωνισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δημόσιες συμβάσεις για εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλειστές de jure και de facto. Η Επιτροπός τα ανέφερε ήδη, πράγματι υπάρχουν προβλήματα και προκλήσεις όταν μιλάμε για την ε, διεθνή διάσταση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα βασικό πρόβλημα για την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές είναι αφενός ε, πολυμερείς ε, συμφωνίες για τις δημόσιες προμήθειες, αλλά και η πρόσβαση στις αγορές ως βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διμερείς συμφωνίες και η ΣΕΤΑ και η ΕΠΑ με την Ιαπωνία είναι επιτυχή παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Τέλος, ειδικά η διεθνής διάσταση έχει την δυνατότητα να προωθήσει την ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Βαλεάν εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, αλλά δεν την βλέπω στην αίθουσα.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 και νομίζω η κατάλληλη στιγμή να τονίσω πως ε, οι τιμές ε, τις οποίες έχουμε ορίσει, τα κατόφλια και στη Γερμανία δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά προκύπτουν από την Παγκόσμια Συμφωνία Δημοσίων Προμηθειών και η γερμανική οικονομία σε αντίθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν σκέφτεται μόνο το Europe First, αλλά θέλουμε να έχουν και οι άλλες αγορές τον ίδιο βαθμό ανοίγματο που επιδεικνύουμε και εμείς. Και θα πρέπει να ασκήσετε, κυρία Επίτροπε, πίεση για να υπάρξει αυτή η αναλογικότητα. Η έκθεση του συναδέλφου Κοέλιο, την οποία χαιρετίζω, νομίζω παρουσιάζει ξεκάθαρα το ότι τελικά δεν υπάρχει λόγος στα κράτη-μέλη ένα 55% των συμβάσεων να δίνεται με βάση τον μειοδότη. Γιατί έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες ήδη από το 2014 για να επιλέγουν οι αρχές τελικά την καλύτερη προσφορά. Γι' αυτό απευθύνω και έκκληση σε όλες τις αναθέτουσες αρχές να σκεφτούν ακριβώς ποιες, ποιους όρους θα βάλουν στις ε, προκηρύξεις για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για να μην παραπονιούνται μετά ότι πάλι κέρδισε ο μειοδότης. Θεωρώ, κυρία Επίτροπε, πως σωστά είπατε ότι με την ψηφιοποίηση στην οποία αποτελεί λαμπρό παράδειγμα η Πορτογαλία μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά ειδικά προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Ντάντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες από το 2014, η Ευρώπη απέκτησε καλή νομοθεσία, των οποίων οι δυνατότητες ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από το μεγαλύτερο μέρος των κρατών μελών η έκθεση, για την οποία ευχαριστώ τον συνάδελφο Κουέλιο και τον δικό μας τον Σκιώδη, τον κύριο Ταραμπέλα, δίνει μια πολύ καλή συνοπτική εικόνα για τη φάση στην οποία έχουν μεταφέρει και εφαρμόσει τους κανόνες τα κράτη-μέλη, αλλά και τα κατεπήγοντα σημεία τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε με την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για την απόδοση των ε, δημοσίων συμβάσεων. Πολύ συχνά πίσω από τη χαμελότερη τιμή υπάρχει αθέμετο ανταγωνισμής και ελάχιστη προσοχή για την βιωσιμότητα και τι κοινωνικέ ανάγκε ή τι περιβαλλοντικέ. Δεύτερον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίες και αυτέ τη ε, κοινωνική οικονομία είναι το 45% τη αξία των συμβάσεων. Αυτό καλύπτουν. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη το πραγματικό του βάρο στην οικονομία. Για το θέμα αυτό θα πρέπει να εγκριθούν ε, συγκεκριμένα δραστικά μέτρα, όπω για παράδειγμα η υποδιέρεση σε παρτίδε τη σύμβαση, εφόσον <coughs> χρειάζεται, ή η εκπαίδευση και κατάρτιση για του εργαζομένου των μικρομεσαίων. Τρίτο, ε, για την οικοδόμηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα πρέπει να αλλάξει και η διαδικασία ψηφιοποίησης της δημόσιας προμήθειας. Θα πρέπει να έχουμε απλουστευμένες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια. Τέλος, να αναφέρω και το θέμα της αμοιβαιότητας των, των δημόσιων συμβάσεων και εκτός Ευρώπης, με τρίτες χώρες. το άνοιγμα των, δημόσιων, των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών μας δεν πρέπει να δυσκολέψει την πρόσβαση των Ευρωπαίων ε, στι αγορέ τρίτων χωρών. Δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη ισορροπία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν λύσει γι' αυτό. Α πούμε με την έγκριση του λεγόμενου εργαλείου για τι διεθνεί δημόσιε συμβάσει, ε, δημόσιε προμήθειε μάλλον, που είναι μπλοκαρισμένο από εσωτερικέ διαπραγματεύσει και αντιρρήσει στο Συμβούλιο. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Μάθιου από του Ευρωπαίου Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστέ, δεν τον βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Επομένως, το λόγο έχει για την ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών ο κύριος Σελίμοβιτς για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Κοέλιο και τους κοιόδης συζήτητες. Οι δυνατότητες ε, των δημοσίων προμηθειών είναι προφανώς πάρα πολύ μεγάλες. 250.000 δημόσιες αρχές ξοδεύουν γύρω στο 14% του ΑΕΠ κάθε χρόνο. 200 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή κάθε χρόνο αγοράζοντας υπηρεσίες και αγαθά. Κι όμως δεν έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως το δυναμικό για τρεις λόγους. Πρώτον γιατί τα κράτη-μέλη καθυστέρησαν στην εφαρμογή της οδηγίας του 2014. Καθυστέρησαν τόσο πολύ ώστε η Κομισιόν έπρεπε να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση κατά κάποιων κρατών μελών και δυστυχώς φοβούμε ότι και πάλι θα καθυστερήσουν στην επόμενη εφαρμογή που αφορά τις ηλεκτρονικές προμήθειες. Δεύτερον, οι αρχές των κρατών μελών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο δεν χρησιμοποιούν τις δημόσιες προμήθειες με τρόπο στρατηγικό. Γι' αυτό τους λέω να μην το θεωρούν ένα διοικητικό βάρος αλλά έναν τρόπο για να προωθηθεί μια έξυπνη και περιεκτική ανάπτυξη για να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες αγορές και νέες θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τρίτον, επειδή οι αρμόδιοι χρειάζονται περαιτέρω κατάρτιση. Είναι κάτι το περίπλοκο αυτό το ζήτημα, οπότε πρέπει να υπάρχει σχετική κατάρτιση και να ε, δούμε ακριβώς ε, τα μαθήματα αυτά στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό καλωσορίζω όλες τις δράσεις που προτείνονται εδώ και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους πάντες πως όλα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει ο κύριος Σόλτες για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα. Συγχαρητήρια, το Άρεστη έκθεση. Όντω έτσι είναι. Οι δημόσιε συμβάσει είναι εργαλείο εξαίρετο για να πετύχουμε διάφορους στόχους. Και ακριβώς, όχι μόνο στο μέτωπο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας και της περιβαλλοντικής πολιτικής, της υγείας, αλλά και ε, των δημογραφικών μεταβαλών. Αυτές οι συμβάσεις έχουν θετικά και αρνητικά. Μίλησαμε για δύο δις που είναι αντικείμενο ε, διαφθοράς. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει γιατί σε κάποιους τομείς οι δημόσιες συμβάσεις κατέληξε να είναι βάρος να είναι πληγή και όχι ατού. Ιδίως όσον αφορά τα είδη διατροφής ε, στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Ε, εκεί θα πρέπει να είμαστε τολμηρότεροι εάν θέλουμε για αυτές τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να έχουμε καλύτερη πολιτική, καλύτερη ποιότητα τροφίμων, ε, λιγότερη διασπάθηση αυτών και έτσι θα βοηθήσουμε και την ύπεθρο. Θα δημιουργήσουμε και τις απασχόλησεις. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα ως αποτελέσματα. Βέβαια προσοχή όσον αφορά την ελάχιστη τιμή, να μην παραβλαβεί η υγεία του κόσμου γιατί η υγεία θα πρέπει να έχει την κορυφαία προτεραιότητα. Άρα, να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά όσον αφορά το φαγητό, τα είδη διατροφής. Θα πρέπει αυτός ο τομέας να εξαιρεθεί. Στην λίστα των ομιλητών, όπως φαίνεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες, ε, δεν αναγράφονται σωστά τα ονόματα με τη σειρά που πρέπει οι τεχνικοί προσπαθούν να ρυθμίσουν το πρόβλημα. Ε, απλώς σας ενημερώνω για να μην παρασυρθείτε σε λάθη. Ε, επόμενος ομιλητής για την ομάδα της αριστεράς είναι ο κύριος Φερέιρα για ένα λεπτό. Mr. Ferreira, you have the floor. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δημόσιες προμήθειες είναι και οφείλουν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο και τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να προασπιστούν και να προωθήσουν τον παραγωγικό του συστό την απασχόληση ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντο μεταξύ άλλων στρατηγικών στόχων. Όμω, μια και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρητικώ ανοίγει, ε, ε, ανοίγει τι πύλε στην ε, μάλλον επιτρέπει να εξεταστούν μόνο εν μέρη κάποιες από αυτές τις ε, προτεραιότητες, είναι πρακτικά δύνατο να ε, αξιοποιηθεί το εργαλείο αυτό, διότι το νομοθετικό πλαίσιο ε, υποχρεώνεται να λάβει υπόψη την υπέρτατη λογική της, του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Δηλαδή η νομοθεσία εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων πολυεθνικών ομήλων που κυριαρχούν στην ενιαία αγορά και αναγκάζουν και μάλλον τώρα έχουν στρέψει την ε, ανεξέλεγκτη όρεξη και απληστία τους στην αγορά των ε, δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να προφυλαχθούν ορισμένοι τομείς, ιδίω οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες, από την όρεξη αυτή, διότι για την ώρα έχουν πληγεί και ιδιωτικοποιηθεί λόγω της δράσης, νομοθεσίας και της πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να μπορέσουν κάποιοι να έχουν κέρδος χάρη στις δημόσιες συμβάσεις. Μπλε κάρτα ο κύριος Βάμπ. Ε, κύριε Σβάμπ, ε, στον κύριο Φερέιρα, ναι. Όχι, σε εσά απευθύνομαι, κύριε Σβάμπ. Επειδή μιλήσατε εκ μέρου τη πολιτική σα ομάδα, θερμή παράκληση είναι να αξιοποιήσουμε τον θεσμό τη μπλε κάρτα για συναδέλφου που δεν έχουν μιλήσει ή δεν πρόκειται να μιλήσουν για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Αν επιμείνετε, οφείλω να ρωτήσω τον κύριο Φερέιρα, αλλά κατευθείαν απευθύνομαι σε εσά. Επιμένετε σε μπλε κάρτα παρότι έχετε μιλήσει. Ωραία. Κύριε Φερέιρα, δέχεστε την μπλε κάρτα. Κύριε Σβάμπ, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Φερέιρα μας είπε ότι φταίνε για όλα οι πολυεθνικές. Γι' αυτό έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, έχετε διαβάσει την νομοθεσία του 2014 και το τι περοβλέπει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερον, τι θέλετε ως επιπλέον κριτήριο επιλογής αν δεν είναι ο ανταγωνισμός. Ίσως έχετε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. You have 30 seconds to answer. 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Αγαπητέ συνάδελφοι, ναι, γνωρίζω το σύνολο της νομοθεσίας που εγκρίθηκε το 2014. Όμως ασχέτως όλων αυτού, με όλες τις ομιλίες που μπορείτε να εκφωνείτε, τα συμφέροντα των πολυεθνικών σίγουρα προστατεύονται όπως με όλα τα νομοθετικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η νομοθεσία σκοπό έχει να μας καθυποτάξει στην λογική του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ενία αγορά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που καταφέρουν να ανταποκριθούν στην ελεύθερο ανταγωνισμό της ενίας αγοράς και ε, καταφέρουν να κυριαρχήσουν. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αυτή η δράση έχει να κάνει και με το πώ έχουν διαλυθεί οι δημόσιε υπηρεσίε σε χώρε όπω τα ταχυδρομεία, σε τομεί όπω τα ταχυδρομεία, η ενέργεια και οι μεταφορέ. Έτσι πλήττονται και οι δημόσιε συμβάσει. Ε, προχωρούμε στον επόμενο μιλητή για την ομάδα Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία, κύριο Άκερ, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δούμε με έναν νέο τρόπο τις δημόσιες προμήθειες έτσι ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων να μένουν τοπικά. Οι παραδοσιακοί κανόνες ε, σημαίνουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, έπαιρναν ε, τις κρατικές συμβάσεις και κατάφερναν να νίκουν τον τοπικό ανταγωνισμό. Στην δική μου την περιοχή, το νότιο ΕΣΕΞ με έκπληξη είδαν ε, οι κάτοικοι πως ο τοπικός πάροχος έχει την έδρα στο Λίβερπουλ, σαν να μην υπήρχε κάποια τοπική εταιρεία. Οι κανόνες λοιπόν πρέπει να αλλάξουν για να σταματήσουν αυτά. Και εδώ πέρα ακριβώς ε, ο Δήμος μου μας δείχνει πώς μπορούμε να το κάνουμε. Προωθεί τα συμβόλαια με βάση την εντοπιότητα και έχουν δείξει οι μελέτες ότι για κάθε λίρα που ξοδεύεται τοπικά 63 ε, πένες παραμένουν στην τοπική οικονομία. Πριν το Πρέστον αλλάξει τις δημόσιες προμήθειες, μόνο μία λίρα στις 20 έμενε στην τοπική οικονομία. Οπωσδήποτε το καλύτερο θα ήταν οι τοπικές λύσεις στις δημόσιες προμήθειες από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι το καλύτερο θα είναι να έχουμε συμβάσεις συντηρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί βεβαίως ε, το κράτος να λέει ότι έχει τελειώσει η κυβέρνησή μας να λέει ότι έχει τελειώσει η λιτότητα, αλλά μπροστά μας έχουμε τρικυμίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας για να μένουν τα λεφτά στις τοπικές επιχειρήσεις. Έχετε μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπίνη. Τη δέχεστε. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφε. Συμφωνώ με αυτό που μόλις είπατε. Όμως, πιστεύετε ότι ίσως οι δημόσιες αγορές ε, από μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις ε, ουσιαστικά κρύβουν μια πονηριά, δηλαδή προσφέρουν χαμηλή τιμή στην αρχή και μετά προσθέτουν ε, με άλλο τρόπο ε, περισσότερα στην τιμή, την τελική που πρέπει να πληρωθεί. Ε, κύριε Άκερ, έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Και εσείς 30 δευτερόλεπτα. Ναι, πολύ σωστό. Ουσιαστικά γίνεται αγώνα προ τα κάτω στο θέμα τη τιμή. Όμω η εμπειρία μα από το Πρεστόν είναι ότι αν κρατήσουμε τι τιμέ ε, τις τιμές στο τοπικό επίπεδο και τι δώσουμε σε τοπικέ επιχειρήσει, οι επενδύσει γίνονται σωστά και απασχολούνται, απασχολούνται περισσότερο μεσοπρόθεσμα ε, οι ντόπιοι. Αυτό στηρίζει και τι τοπικέ κυβερνήσει. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κι εσεί. Καλό θα ήταν να αλλάξουν τα πράγματα για να μπορέσουν να μείνουν τα κονδύλια στο τοπικό επίπεδο και να βοηθήσουμε τι τοπικέ οικονομίε. Να επαναλάβω προς τους συναδέλφους ότι οι ηλεκτρονικοί πίνακες λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν εμφανίζουν τη σωστή σειρά των ομιλητών. Κατά συνέπεια, μέχρι ότου οι τεχνικοί να διορθώσουν το πρόβλημα, ε, να μην τους παίρνετε υπόψη. Ε, επόμενη ομιλήτρια για την ομάδα των Εθνών και της Ελευθερίας, η κυρία Τροτσίνσκι για ένα λεπτό. Πρόκειται για σεβασμό κάποιε διοντολογίε όταν έχουμε αυτέ τι δημόσιες Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα έπρεπε να χρειάζεται αυτό το κείμενο. Είναι κάτι αυτονόητο, λογικό. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα το, η προϋπόθεση της διαφάνειας και υπάρχουν και, και άλλες αρχές οι οποίε είναι αδιαπραγμάτευτε. Είναι πρόβλημα τι γίνεται με τι τρίτε χώρε όσον αφορά την ειδική κυριαρχία, την ανεξαρτησία. Οπότε θα έπρεπε ανεξάρτητα να θεσπίζονται κάποια κριτήρια για τι ε, επιχειρήσει, οι οποίε συμμετέχουν και κερδίζουν αυτού του διαγωνισμού, οπότε θα πρέπει να δούμε ότι μεταξύ των ε, πιο εθνικιστών και των φιλελευθέρων ε, μια διαφορά. Εμεί θεωρούμε το περιβάλλον και η κοινωνική πολιτική είναι το πιο βασικό. Δεν θα πρέπει να γνωρίζει σύνορα αυτό το όραμα. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα, τα όρια των δυνατοτήτων μας, γιατί πρόκειται για ε, θέμα εθνική προτίμηση και γι' αυτό είμαστε κατά αυτού του κειμένου. Των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, το λόγο έχει ο κύριος Σονιέρτς, μη εγγεγραμμένος. Trudno słuchać tych e, opowieści o tym, jak to e, zamówienia publiczne są. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω και από ό,τι φαίνεται οι δημόσιε προμήθειε είναι το κέρας της αμάλθειας. Όχι ακριβώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εξοδεύουν τα λεφτά των άλλων. Όχι, δεν είναι σωστό. Το σωστότερο είναι να εξοδεύει κανεί τα λεφτά του, τα δικά του, σε πράγματα τα οποία χρειάζεται ο ίδιο. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, πρέπει να αποσυρθεί το κράτος από όλους τους τομεί όπου δεν χρειάζεται. Και έτσι δεν θα έχουμε πλέον ε, ανέντιμους ε, υπαλλήλους. Λοιπόν, αν ε, βασίζεται από την άλλη κανείς στο κριτήριο του μειοδότη, είναι κάτι το οποίο επαληθεύεται εύκολα. Αν μπούμε σε κοινωνικά κριτήρια, θα ε, καταλήξουμε σε ένα μόνο άτομο που πληρεί όλα τα κριτήρια, τον υπάλληλο ο οποίος ε, παίρνει την απόφαση. Πρέπει λοιπόν να αποσυρθεί το κράτος. Νίμπλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα σημείο θα ήθελα να τονίσω από την εξαιρετική έκθεση Κοέλιο, το οποίο θεωρώ σημαντικό. Αναφέρεται στην έκθεση ότι ο αριθμός των προκηρύξεων με μία μόνο προσφορά από το 2006 μέχρι το 2016 ανέβηκε από το 14% στο 29%. Δηλαδή ένα τρίτο των διαγωνισμών έχουν μία μόνο προσφορά. Ε, είναι πολύ ανησυχητικό νούμερο αυτό. Αν ε, δούμε τις αιτίε, ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύς κόπος να ε, λάβουν μέρος και να υποβάλουν προσφορά. Στην ε, δική μου την πόλη φτιάξαμε ένα νέο σχολείο, ξεπερνούσε το κατόφλι των 5 εκατομμυρίων, άρα κάναμε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, αλλά πάλι το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το διοικητικό άχθος και τελικά υπάρχει μία μόνο προσφορά. Τι θέλω να πω. Ε, θέλω να τονίσω αφενός ότι στις ε, δημόσιες προμήθειες ε, πρέπει να δούμε και το διοικητικό βάρος και στην επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να δούμε τους κανόνες ε, περί δημοσίων προμηθειών, ειδικά το θέμα των χρηματικών ορίων των κατοφλιών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν είναι δυνατόν μετά το 1 τρίτο των ε, διαγωνισμών να έχουν μία και μόνο προσφορά. Άρα κάτι πρέπει να διορθωθεί εδώ πέρα γιατί δεν έχει κάποιο νόημα στην ε, Βαβαρία παραδείγματο χάρη ε, να ζητούμε πρόσφορες για τα σχολεία από την Κύπρο ή την Πορτογαλία κτλ. Το λόγο έχει η κυρία Ροζιέρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή μας, τον κύριο Ταραμπελά, για τη δουλειά του. Υπόθηκε του θυμίσατε του αριθμού. Γνωρίζουμε ότι 14% του ΑΕΠ, 12 δις ευρώ το χρόνο, είναι η αξία των δημόσιων ε, προμηθειών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι σημαντικό λοιπόν για να μεταφράσουμε την, ε, τις δημόσιες επενδύσεις σε κάτι άλλο από απλό πολλαπλασιασμό του κέρδους των πολυεθνικών. Η νομοθεσία όμως το 2014 δεν αξιοποιείται ακόμη από τους ε, δημόσιους αγοραστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, η ε, διαλλακτικότητα που προτείνει η δηληξία για να χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια από τη χαμηλότερη τιμή ε, στοιχεία όπως η κοινωνική συμμετοχή, η περιβαλλοντική προστασία στην εξέταση των προσφορών είναι κριτήρια που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν οι δημόσιοι αγοραστές, οι αναθέτουσες αρχές να αναλάβουν δράση για να υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα ενάρτη και Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δημοσίες προμήθειε είναι μια πολύ ευαίσθητη δραστηριότητα όπου το κράτος πρέπει να επιδείξει ότι πραγματικά ξοδεύει προσεκτικά τα χρήματα των φορολογουμένων. Αφενός πρέπει να υπάρχει τάξη και αφετέρου πρέπει να υπάρχει ακριβώς εξοικονόμηση. Και πρέπει να υπάρχει και η διαφάνεια για να ξέρει ο κόσμος τι κάνει το κράτος με τα λεφτά του. Οπότε οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να παρακολουθήσει τι σημαίνει. Ταυτόχρονα εδώ θα επιτύχουμε μόνο εάν οι διαδικασίες αυτές δεν είναι γραφειοκρατικές. Όπως είπε και η κυρία Νίμπλερ, δεν μπορούν να μπαίνουν όλα εδώ στο ίδιο καζάνι. Αλλιώς ε, θα έχουμε θεωρητικά πολύ ωραίους κανόνες, αλλά στην πράξη δεν θα εφαρμόζεται τίποτα, γιατί οι εταιρείε δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους όρους. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μήπως σε κάποιους τομείς να αλλάξουν τα κατόφλια για να μην παράγουμε μόνο αχρίαστη γραφειοκρατία. Mr. you have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Αναγνωρίζουμε νομίζω ότι είχαμε την οδηγία του 2014 η οποία ήταν μια βελτίωση γιατί δεν κοιτάμε μόνο τις τιμές αλλά και την ποιότητα. Βεβαίως αυτό μας οδήγησε σε κάποια προβλήματα στην Ολλανδία γιατί οι περισσότερες προμήθειες γίνονται σε επίπεδο Δήμου και όταν μιλάμε ακριβώς για την παροχή φροντίδας ε, σε άτομα τα οποία την χρειάζονται. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία ακριβώς για να ανταποκριθούν στους κανόνες του 2014 και ε, αυτό προέκυψε από μια κομισιόν η οποία μας λέει ότι έχει ως στόχο την καλύτερη νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε κύριε Πίτροπε σε δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα είστε διατεθειμένοι να δώσετε περισσότερο περιθώριο στα κράτη-μέλη για να μην υφίστανται ακριβώς τις αρνητικέ συνέπειες αυτής τη νομοθεσίας στον τομέα τη τοπικής παροχής φροντίδας και δεύτερον έχετε δει τι αποτέλεσμα έχει αυτή η νομοθεσία ακριβώς σε αυτόν τον τομέα και στις μικρομεσαίες Η είδηση για τους συναδέλφους, η ακρίβεια αυτών που γράφουν οι ηλεκτρονικοί πίνακες για τη σειρά των ομιλητών αποκαταστάθηκε. Επόμενο ομιλητής θα έπρεπε να είναι ο κύριο Πρέτσελ. Δυστυχώ, ούτε αυτό είναι στην αίθουσα. Κάτι περίεργο συμβαίνει σήμερα, αρκετέ απουσίες. Επομένως, τον λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ζαριανόπουλος. Οι δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή η ιδιωτική εκμετάλλευση δημόσιας περιουσίας, αποτελούν τεράστια αγορά, πεδίο κερδοφορίας τρισεκατομμυρίων και ανταγωνισμού των μονοπωλίων σε ευρωνησιακό και παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια θερμοκήπιο σκανδάλων γι' αυτό και η ανησυχία και η επιθετική στρατηγική της ένωσης για διασυνοριακό άνοιγμα συμβάσεων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών αλλά και προστατευτισμού της απέναντι στις τελευταίες ακόμα και με προσαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης στα μονοπωλιακά συμφέροντα. στην ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις δημόσιες συμβάσεις με ιδιώτες σημαίνει τσουνάμι fast track ιδιωτικοποιήσεων των πάντων. παραδόθηκαν δρόμοι αεροδρόμια λιμάνια ακτοπλοεία συγκοινωνίε, ορυκτός πλούτος ενέργεια τηλεπικοινωνίες το νερό βουνά παραλίες στρατιωτικές παραγωγικές υποδομές υδρογονάνθρακες ανακύκλωση υγεία παιδεία τα πάντα. αποκορύφωμα η παράδοση όλης της δημόσιας περιουσίας της χώρας για 99 χρόνια από την κυβέρνηση σύριζα ανέλθους δανειστές. φυσικός πλούτος και πλούτος βγαλμένος από τους φόρους και τον ιδρώτα του λαού καλεί το ίδιο να τον ξαναπληρώσει στα ταμεία των ιδιωτών με διόδια αύξηση τιμολογίων δάνεια και ευρωνοσιακές επιδοτήσεις που φορτώνεται μόνος δρόμος να βγει από τη μιζέρια να ικανοποιήσει τις ανάγκες του όλος αυτός ο πλούτος να γίνει λαϊκή περιουσία με κεντρικό σχεδιασμό εργατικό έλεγχο και λαϊκή εξουσία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σάινφελτ για δύο λεπτά. E, e, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο από πλευράς απασχόλησης αλλά είναι και σημαντικό γιατί εδώ μιλούμε για μεγάλα χρηματικά ποσά. Ε, θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί ότι για το 2014 αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σημεία έχουμε στα κριτήρια μόνο την τιμή. Θα έπρεπε να έχουμε και ποιοτικά κριτήρια επίσης. Επίσης, να μην ξεχνούμε τον κύκλο ζωής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Μην σκεφτόμαστε μόνο την πρώτη φάση. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη το ρυθμό των εξελίξεων, οπότε έχουμε να κάνουμε με τέτοια προϊόντα. Ε, γιατί νομίζω ότι με τις δημόσιες συμβάσεις τονώνεται η τεχνολογική πρόοδος. Να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία και να δώσουμε στην υπόθεση αυτή περισσότερη ευελιξία. Οι εταιρείε θα πρέπει να προσαρμοστούν στις αλλαγές που Τώρα βέβαια το κόστος των εργατικών είναι ευξημένο και θα πρέπει να βρούμε τρόπο για περισσότερη ευελιξία γιατί ξέρετε πάρα πολλέ εταιρείε τελικά παρετούνται δεν μπαίνουν στον χώρο του ανταγωνισμού για να κερδίσω κάποιους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μίτση για ένα λεπτό. Μικρό, please. μικρόφωνο σας, λέει ο πρόεδρος, στην κυρία Μίτση. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση αντιστοιχεί σε μια στρατηγική. Πρέπει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα ούτω ώστε οι δημόσιοι αυτοί διαγωνισμοί και αυτές οι προμήθειες να πηγαίνουν χέρι-χέρι με την πρώτη τεχνολογία, να έχουμε μια στρατηγική που να είναι πιο προσβάσιμη στον κόσμο, στις κυβερνήσεις αλλά και στις εταιρείε. Πολύ σημαντική επομένως η έκθεση. Έτσι θεσπίζεται ένα τέτοιο σύστημα ηλεκτρονικό. Υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και έτσι δημιουργείται η σχετική πλατφόρμα. Οπότε έτσι τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να εφαρμοστεί σωστά ε, αυτό το κείμενο. Εμείς ήδη έχουμε νομοθεσία για αυτές τις δημόσιες συμβάσεις. Το, αποκτήσαμε αυτή την νομοθεσία πολύ νωρίς, πιο νωρίς από όλα τη μέλη. Ε, βέβαια και εμείς για λόγους διαφάνειας θα συμμορφωθούμε. Οι δημόσιες συμβάσεις, ειδικά σε ορισμένα κράτη-μέλη, αποτελούν χρονίουσα πληγή και πηγή διαφθοράς δυστυχώ όμω έχουν υπάρξει περιπτώσει στι οποίε και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν είχαν και την καλύτερη διαγωγή. είναι θεμητή η εξέβρεση νέων μεθόδων ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και βελτιστοποίηση των υφισταμένων με γνώμονα πάντα τη μεγαλύτερη διαφάνεια τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία για το δημόσιο συμφέρον. προσωπικά όμω θεωρώ πω η χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να εξακολουθήσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάθεση συμβάσεων με την παράλληλη εισαγωγή νέων κριτηρίων. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην παραβιάζει την κυριαρχία των κρατών μελών τα οποία και πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο σε κάθε δημόσια σύμβαση. ταυτόχρονα όμω πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι διαγωνισμοί ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα εκτεταμένη διαφθορά όπω έχουν παρατηρηθεί σε πολλέ χώρε τη ενώσεω. βασικό σκοπό πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα η πάταξη τέτοιων φαινομένων. δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε σε ορισμένου να πλουτίζουν ει βάρο των πολιτών. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γκραπίν για ένα λεπτό. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ καλό που έχουμε έκθεση του Κοινοβουλίου μας για το θέμα αυτό. Και είναι πολύ θετικό να ξαναδούμε το όλο ε, θέμα της νομοθεσίας του 2014 για τις δημόσιες προμήθειες. Τότε, άλλωστε, δεν ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τι οδηγίε που είχαν εγκριθεί και να γιατί βλέπουμε ότι είχα δίκιο. Η οδηγία ήταν αρκετά γενικόλογη. Άφηνε πολύ περιθώριο να συνεχίσουν να υπάρχουν σοβαρέ ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών για τι εθνικέ του στρατηγικέ για τι δημόσιε προμήθειε. Τώρα δεν είναι ξεκάθαρο πώ μπορούν κάποια πράγματα να διευθετηθούν, όπω ε, προσφυγέ, τα παράπονα γίνονται πολύ μεγαλύτερες ε, οι προθεσμίες και διαρκούν πολύ διαδικασίες ώστε καθυστερούν και επενδύσεις ή για το ποιο μπορεί να υποβάλει, να κάνει μια προσφυγή. Ένα κατάστημα δεν μπορεί να κάνει ε, προσφυγή για υποδομές αυτοκινητοδρόμου ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι το 60% των αγορών δεν γίνονται μόνο με την καλύτερη τιμή. Και για την έρευνα, στο ενωτρικό τομέα ας πούμε, αυτός ο τομέας θα πρέπει να αποκλείεται από τις δημόσιες προμήθειες στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Έχω δεχθεί 7 αιτήματα. Τα κάνω και τα 7 αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Ντόρφμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν εισηγητής ε, για την γνωμοδότηση στην ΕΝΒΗ και στην έκθεσή μου εστιάστηκα κυρίως στην προμήθεια τροφίμων από τον ε, δημόσιο τομέα, παραδείγματος χάρη σε σχολεία, και νοσοκομεία. Θεωρώ ότι ακριβώς εκεί οι πελάτες αλλά και οι ε, γονείς των μαθητών επιθυμούν τοπικά τρόφιμα και θα είναι παράλογο να υποχρεώνονται να αγοράζουν ε, ε, τρόφιμα κατόπιν πανευρωπαϊκής προκήρυξης. Αντιλαμβάνομαι την εσωτερική αγορά, αλλά νομίζω ότι για τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των πελατών, των χρηστών δηλαδή. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στην προκήρυξη να προτιμούνται τοπικά τρόφιμα. Το λόγο έχει ο κύριος Πάλμερ για ένα λεπτό. Παρακαλώ το κοινό σύμφωνα με τους uh, κανονισμούς δεν επιτρέπεται να χειροκροτά. Μπορεί να ακούει, να σκέφτεται, αλλά όχι να παρεμβαίνει με χειροκροτήματα. Ο κύριος Πάλμερ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα οποία ακούστηκαν για την ανάγκη να γίνουν οι προμήθειες πιο προσβάσιμες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως να μίσω συγκεκριμένα είναι το σκάνδαλο της σύγχρονης δουλείας που αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην χώρα μου 136.000 ε, άτομα υπολογίζεται ότι έχουν πέσει θύμα της σύγχρονης δουλείας του 2017. Θα ήταν σκάνδαλο εάν ε, η ε, δουλεία αυτή στηρίζεται μέσω δημοσίων κονδυλίων, μέσω των δημοσίων προμηθειών. Οπότε, εγώ υποστηρίζω και ελπίζω να με στηρίξει το Κοινοβούλιο κάποια δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα μέσω των προμηθειών. Παραδείγματο χάρη να υπάρξει μια χάρτα κατά τη σύγχρονη δουλεία όπως αυτή που υπογράφουν οι Δήμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται αυτή η πρακτική έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο για αυτό το σημαντικό θέμα. Σε ό,τι αφορά τι κρατικέ προμήθειε, οι μεγάλε φαίνεται να συμφέρουν όλε. Οι μεγάλε εταιρείε, οι μεγάλε επιχειρήσει αγαπιούνται από του περισσότερε αναθέτησε αρχέ. Όμω και το μικρό μπορεί να είναι όμορφο. Οι μικρέ εταιρείε μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικέ, πιο αποδοτικέ και πολλέ φορέ και φτηνότερε. Δυστυχώ όμω οι μικρότερε εταιρείε πολλέ φορέ αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε δημόσιου διαγωνισμού. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που μπορώ να εγκρίνω την ε, έκθεση αυτή που σκοπό έχει να αποκαταστήσει αυτή την κατάσταση. Πρέπει όμω να πάμε μακρύτερα. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια, μικρότερε εταιρείε πλήττονται από τι καθυστερημένε πληρωμέ, από τι περιχοκλάδε τη γραφειοκρατία και από τη γραφειοκρατική τεμάχηση των ε, υπηρεσιών τι οποίε πρέπει να υπερπηδήσουν για να μπορέσουν να υποβάλουν ό,τι χρειάζεται αφού κάνουν τη δουλειά του. Οι μικρέ εταιρείε λοιπόν είναι καλέ, είναι η καλύτερη λύση για τι κυβερνήσει και για του τοπικού εργαζομένου. Πρέπει να τι ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ. Λόγο έχει ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάθε κράτο συνάπτει ένα διαμοιβή συμβάσει με διάφορε εταιρείε και εγχώριε και εταιρείε του εξωτερικού οι συμβάσει αυτέ παίζουν ε, σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη τη οικονομία του κράτου ε, διότι συνήθω γίνονται σε τομεί με μεγάλη στρατηγική σημασία όπω είναι η βαριά βιομηχανία τα δημόσια έργα οι κατασκευέ η ενέργεια οι τηλεπικοινωνίε και άλλα. με τι συμβάσει λοιπόν αυτέ το κράτο προσπαθεί να προωθήσει την οικονομική και όχι μόνο πολιτική του αρκεί βεβαίω να μην έχει εκχωρήσει όλε τι παραγωγικέ του πηγέ στου ξένου όπω έχουν κάνει οι τελευταίε κυβερνήσει στην ελλάδα λόγω τη εφαρμογή των μνημονίων. εν πάση περιπτώσει ε, για να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθεια εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει δυνατότητα προσβάσεως και σε αγορές τρίτων χωρών. Ε, οι χώρες αυτές έχουν ε, λόγω προστατευτισμού δημιουργήσει δυσχέρειες στην πρόσβαση και στις προσφορές από εταιρείες ευρωπαϊκές. γι' αυτό λοιπόν το λόγο και για να υπάρχει μια ισορροπία στα μέτρα του θεμητού ανταγωνισμού θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι ευρωπαϊκές χώρες τις ε, οδηγίες που έχουν δοθεί με την ε, ε, μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις συμβάσεις. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χέτμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δημόσιες συμβάσεις και η νομοθεσία που τις διέπει είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση για τη κοινωνία σε κάθε επίπεδο. Μπράβο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και μπράβο για αυτές τις έξι ε, προτεραιότητες τις οποίες ανέδειξε. Θα πρέπει αυτές οι συμβάσεις να διέπονται από ε, σαφήνεια και επίσης τα σχετικά να είναι κατανοητά. Άρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρονικές τέτοιες ε, συμβάσεις και διαγωνισμούς. Να μπορούν όλα να γίνονται ιντερνετικά. Βεβαίω και χρειάζεται να δούμε καλύτερα τα κριτήρια ε, για την ε, κατακύρωση και να μην έχουμε μοναδικό κριτήριο την τιμή. Το λόγο έχει ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 250.000 δημόσιοι φορείς αναθέτουν ε, δημόσιες συμβάσεις για έργα για προμήθειες για υπηρεσίες. το κόστος είναι δύο εκατομμύρια ευρώ το 14% του αεπ. αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για τεράστια για σημαντικά ποσά των φορολογουμένων και φυσικά έχει αποδειχθεί ότι στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων επί της ουσίας έχουν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα ταυτόχρονα οι δημόσιε συμβάσει θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη να δημιουργήσουν θέσεις εργασία, να συμβάλλουν στην ενίσχυση τη στρατηγική του ίδιου του κράτου, λαμβάνοντα υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει έχουν πάρει μόνο το 45 των αναθέσεων ενώ το 55 των αναθέσεων έχουν πάει με βάση την αρχή τη χαμηλή τιμή, δηλαδή του μειοδότη που δεν σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχει μια εγγύηση ότι τα έργα είναι αποδοτικά. ταυτόχρονα η διεθνοποίηση είναι αυτή η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ευρωπαϊκή ένωση καθώς ανοίγει την αγορά όπως έγινε με την σύμβαση της ceta ή της ttip ενώ άλλες τρίτες χώρες κρατούν κλειστές τις δικές τους αγορές ας εξετάσουμε λοιπόν ορισμένα στοιχεία είτε την τοπικότητα είτε την εθνική προτίμηση ως στοιχεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σδρογεύσκη για ένα λεπτό ολοκληρώνει την διαδικασία του Catch ε, przyznam, że jestem zwolennikiem ograniczania ilości środków finansowych. Ευχαριστώ να σας ομολογήσω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές στο πόσα ξοδεύει ο δημόσιος κορδοβανάς για αυτές τις συμβάσεις. Δεν είμαι υπέρ του να έχουμε θεσμικά όργανα όπως τις τοπικές αρχές που να έχουν τέτοιου είδους αρμοδιότητες, τέτοιου είδους οικονομική δραστηριότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος σε τέτοιους φορείς. Βέβαια, μπράβο στον κύριο Κοέλιο γιατί τα πήγε πολύ καλά με αυτή την έκθεση και διαπιστώσαμε ε, τα εξή δύο που αφορούν την ποιότητα των διαγωνισμών. Πρώτα-πρώτα ένα εξωτερικό πλαίσιο. Αυτό είναι η νομοθεσία. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχει ακρίβεια όσον αφορά την ακολουθητή διαδικασία. Ε, για αυτό το δεύτερο δυσκολευόμαστε ιδιαίτερως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε για τη διαδικασία του Catch the Εξ ονόματος της Επιτροπής, το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Μπιανκόφσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη συζήτηση φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και θέλω και πάλι να επαναλάβω ότι ο λόγος που αποφασίσαμε να εγκρίνουμε το πακέτο αυτό, τη δέσμευτη μέτρων, δεν είναι γιατί η νομοθεσία μα είναι κακή. Η νομοθεσία είναι ολοκένουργια, είναι και φρεσκότατη, αλλά από την πλευρά μα πιστεύουμε ότι η νομοθεσία αυτή, παρόλο που είναι καλή, έχει κακή υλοποίηση. Η νομοθεσία που πολλοί σχολιάσατε ότι δεν προβλέπει αρκετή ελαστικότητα, η διαλεκτικότητα για την εφαρμογή των κανόνων, επιτρέπει μεγάλο περιθώριο. Βεβαίως πρέπει να, να τηρεί τον νόμος. Όμως, για τις κοινωνικές υπηρεσίες πούμε, προβλέπει πολλά. Αφήνει πολύ περιθώριο. Δίνει τη δυνατότητα ενός υπιότερου συστήματος για να ενσωματωθούν όλα τα κοινωνικά κριτήρια εφόσον κάποιος θέλει στους δημόσιους διαγωνισμούς. Οπότε για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα ετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν. Επίσης συμφωνούμε ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων προμηθειών είναι εξαιρετικά σημαντική αποτιμία γιατί θα συμβάλλει κατά την άποψή μας στο να βελτιωθεί η διαφάνεια, ιδίω για τις καθυστερημένες πληρωμές και μετά οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε αύξηση. Είδαμε ότι στα κράτη-μέλη που ε, εφαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικέ δημόσιε συμβάσει, δημόσιε προμηθείε, αυξήθηκε η συμμετοχή των μικρομεσαίων. Βεβαίω, είναι μόνο λίγα ακόμη τα κράτη-μέλη που έχουν ε, προβλέψει τέτοια δυνατότητα. Όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει για όλο τον κύκλο εργασία και δράση των δημόσιων προμηθειών να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακή συμμετοχή. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολλές προσωπικές ε, γνώσεις για το θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι σοβαρό το βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξέρετε αυτή η νομοθεσία που προτείνεται. Είναι τελείως ε, ένα Είναι μια ε, λύση είναι μια μάλλον ε, εντύπωση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η εταιρική σχέση που επιζητούμε δεν απαιτεί αλλαγή της νομοθεσίας. Κάποιες κατευθυντήριες γραμμές απαιτεί, κάποιες συστάσεις. Κάποιοι φοβούνται ότι θα παρεμποδιστούν από το να λάβουν τη σωστή απόφαση γιατί δεν έχουν αρκετές ικανότητες ή δεξιότητες. Δεν είναι έτσι. Η καθυστερημένη επίσης μεταφορά ε, της οδηγίας οφείλεται και στην έλλειψη στατιστικών δεδομένων. Α πούμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στη Γερμανία, διότι η μεταφορά έχει αργήσει πάρα πολύ στα κρατήδια. Δεν ξέρουμε πώ ακριβώ έχουν πάει τα πράγματα στην πράξη. Απλώ να προσθέσω ότι από την έγκριση έχουμε και εξάντα εργαλεία για τα μεγάλα ε, προγράμματα και έργα για να βοηθηθούν οι τέτοιο αρχές και οι αγοραστέ να αποφύγουν προβλήματα ενώ οργανώνουν διαγωνισμού και διαθέτουν μεγάλα ποσά για προγράμματα. Έχουμε φροντίσει να δημοσιευτούν εκατοντάδε συστάσει για τα επαγγελματικά προσόντα. Υπάρχουν και σχετικέ συστάσει, αλλά όπω είπα, ο επόμενο γύρο θα είναι για τι κοινωνικέ δημόσιε προμήθειε. Ε, έχω λοιπόν τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και για τους στόχους μας και θέλω η συζήτησή μας να παραμένει ζωντανή γιατί το θέμα αυτό το αξίζει. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με τον εισηγητή κύριο Κοέλιο, ο οποίος έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο Μπιενκόφσκι για τα σχόλιά της. Όπως είπατε κι εσείς, Έχουμε ε, μπροστά μας μια ξεκάθαρη περίπτωση όπου η Ευρώπη έκανε κάτι καλό, εμείς εγκρίναμε εγκαίρως το νομοθετικό μας πλαίσιο και τα προβλήματα προκύπτουν από την βραδεία και κάποιες φορές εσφαλμένη υλοποίηση από την πλευρά των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα από τους εαυτούς μας, θα πρέπει τα κάτι μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάψουν να ε, καταστρέφουν αυτό που φτιάξαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι ε, συνεισφορέ του και να τονίσω τρία σημεία. Πρώτον, νομίζω ότι υπάρχει γενικώ συνένεση σε σχέση με του ε, απότερου στόχου τη πρωτοβουλία αυτή. Την ιδέα ότι με το εργαλείο αυτό μπορούμε να προβλέψουμε περισσότερη διαφάνεια για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό και να έχουμε εργαλεία για να επιδιώξουμε στόχους καινοτομίας, οικολογικής και κοινωνικής ε, οικονομίας, βιώσιμης και συμμετοχικής ανάπτυξης. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Νομίζω ότι ε, γενικώ στι παρεμβάσει ακούστηκε ότι χρειάζονται στήριξη. Και τρίτον και τελευταίο, η ιδέα της ψηφιοποίησης. Δεν αρκεί ένα απλό εργαλείο για την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά σημαντικό είναι να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια με την ψηφιοποίηση. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους, κύριε Πρόεδρε. οι συνεισφορές τους θα ληφθούν υπόψη και είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι την εμπιστοσύνη μας, αυτή που μας δείχνουν οι πολίτες, θα την εκφράσουμε και με τις συστάσεις που θα εγκρίνουμε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η πρώτη συζήτηση έχει ως θέμα επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του χάρτη 97. Δίνω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Τάνοκ εκ των συντακτών της ερώτησης. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω με κάποια επιφύλαξη με κάποια επιφύλαξη την απόφαση του 2016 για χαλάρωση κάποιων ε, κυρώσεων εις βάρος της Λευκορωσίας. Αλλά τώρα, δεδομένης της προσάρτησης της ε, Κρυμαίας από την ε, Ρουσία, και την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία υπάρχει αίσθηση ότι ο Λουκασένκο μπορεί να ε, θέλει θερμότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντισταθμίσει την ρωσική επιρροή φοβούμενος ότι μπορεί και αυτός να βρεθεί στην θέση της Ουκρανίας και του Γιανουκόβιτς Μπορεί έτσι να έχουμε αποτελέσματα για μεγαλύτερη ελευθερία και για να ανοίξει η χώρα στην ε, Δύση. Όμως, όπως βλέπουμε με την ε, χάρτα του 97 όλα αυτά ήταν πολύ αισιόδοξα. Βλέπουμε ότι υπάρχει στοχευμένη δίωξη δημοσιογράφων, ε, απειλές για την ζωή τους όπως στην περίπτωση της κυρίας Σαραντίνα. Οι ελπίδες του να αλλάξει στάση ο Λουκασέγκο ήταν προώρες. Θα πρέπει λοιπόν ε, κάποια στιγμή να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας. Λόγο έχει ο κύριος Αουστρεβίτσιους για ένα λεπτό επίσης εκ των συντακτών της ερώτησης. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα μιλάμε για την ελευθερία του τύπου ή την απουσία της στην Λευκορωσία. Στοχεύουν το διαδίκτυο. Όλοι όσοι σχολιάζουν στο διαδίκτυο θα πρέπει να καταγραφούν και τα δεδομένα τους να μεταφέρονται στην KGB. Η ΚΑΓΚΕΜΠΕ έχει όπως ξέρετε ε, ανεξάντλητη φαντασία και εξουσίες. Πρέπει λοιπόν δεν αρκεί απλά να επαναλάβουμε τις ανησυχίες μας για την ιστοσελίδα χάρτης 97 θα πρέπει να αρθεί το μπλοκάρισμα της ιστοσελίδας να στηριχθεί οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ο Λουκασένκο το τέρας αυτό δημιουργεί ένα πυρηνικό τέρας ε, το εργοστάσιο ενέργειας στο Αστρεβίτς που θα υπονομεύσει τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες ε, των Λευκορώσων και ολόκληρη της Ευρώπης ε, στο δικαίωμα στην ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να θέσουμε αυστηρούς όρους. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής πρέπει να σταματήσουν να είναι αφελείς. Δεν παριστάνει καν ότι αλλάζει το Μίνσκ. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να σταματήσουμε αμέσως τις διαπραγματεύσεις και να κάνουμε κάτι σοβαρό. Θα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητή συνάδελφοι, η Λευκορωσία σήμερα είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει ξεκάθαρα το πόσο ο περιορισμός των ΜΜΕ και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια της χώρας, της περιοχής και ολόκληρης της Η Λευκορωσία επέζησε μία εκ των μεγαλύτερων πυρηνικών καταστροφών στην ιστορία και τώρα ξανασχολείται με τα πυρηνικά, μια περιπέτεια που μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση χειρότερα από το Τσέρνομπιλ. Η Λευκορωσία έχει περιορίσει τα ανεξάρτητα ΜΜΕ όπως τον χάρτη 97. Ταυτόχρονα έχει επιτρέψει στο καθεστώς του Πούτιν να φτιάξει ένα πυρηνικό τέρας στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και η Σοβιετική Ένωση είχε αναστείλει την οικοδόμηση αυτού του πυρηνικού εργοστασίου μετά του Τσερνομπίλ. Με ρωτάνε συνεχώς οι πολίτες μου τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά. Ερωτώ την Κομισιόν πώς θα διασφαλίσουμε ακριβώς αυτό το τον έλεγχο του πυρηνικού εργοστασίου. στην Λευκορωσία δίνουμε εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων μας και χρησιμοποιούνται τελικά για κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων και κατάπνιξη των Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι θεμελιώδης ευρωπαϊκή αξία και πρέπει να διαφυλάσσεται. Θα πρέπει να είναι και ένα απόσπαστο τμήμα των σχέσεων της Ένωση με την Λευκορωσία. Ο χάρτη 97 είναι ένα παράδειγμα για το πώς οι αξίες μας υπονομεύονται. Αυτό το ειδησιογραφικό ε, στότοπο ε, έκλεισε στη Λευκορωσία, απαγορεύτηκε και η αρχιστάκτρια φυλακίστηκε σε προσπάθεια να θυμωθεί η φωνή του κοινού. Άλλε ιστοσελίδε και μέσα επίση διώκονται για να μην υπάρχει ελευθερία του λόγου με την ε, ανωνυμίας. Αυτή είναι μια ανησυχητική τάση μιας ε, υπονόμευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ένα περιβάλλον καταπίεσης. Η Λευκορωσία δεν επιτρέπει και την ελευθερία του να θρίζεστε. Με ε, επίθεση σε ανεξάρτητους ε, συνδικαλιστές. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε τις περισσότερες κυρώσεις που βάριναν τι λευκορωσικέ επιχειρήσει και του επιχειρηματίε. Σε πνεύμα συμφιλίωση, ελπίζοντα ότι οι καλύτερε σχέσει θα οδηγούσαν σε περισσότερο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Τώρα είναι σαφέ ότι αυτό δεν έδωσε αποτελέσματα. Η περίπτωση του Χάρτη 97 και ορισμένων ε, συνδικαλιστών έκαναν αυτή την περίπτωση τελείω ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή η ΕΕ θα πρέπει να προβλέψει χρηματοδότηση για τέτοιες ε, για τέτοιους ε, ε, οργανισμούς όπως η Μπέλτα και ο Χάρτες 97. Θα πρέπει να υποστηριχθούν και να υπάρξει άμεση δράση και βοήθεια. Η στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λευκορωσία πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένου όρου και προποθέσει. Και θα πρέπει να υπάρχουν και συνέπειε όταν αυτέ οι προποθέσει δεν πληρούνται. Η παρενόχληση, οι απειλέ κατά τη ζωή, η φυλάκιση δημοσιογράφων και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδικαλιστών και άλλων είναι οπωσδήποτε παραβιάσει που θα πρέπει να κοστίσουν στη Λευκορωσία τη χρηματική τη υποστήριξη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ούρμπαν Κρέσπο για 1,5 λεπτό. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά έχουμε να κάνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά που έχουμε το Κοινοβούλιο γιατί εδώ αναδεικνύεται η καταστολή στη χώρα και βλέπουμε ότι έτσι εμποδίζεται πιο μεγάλη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο μεγάλη δημοκρατική συμμετοχή του κόσμου εκεί. Όμως το 2014 μέχρι το 2017 είχαμε αυτό το πακέτο ενίσχυσης προς τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έφτασε στα 91,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε μια συμφωνία για την κινητικότητα των φυσικών προσώπων, φοβερή σύμπτωση. Όλα αυτά τελικά ήταν για να ε, γίνουν στρατόπεδα για τους μετανάστες. Δηλαδή να γνωρίζουμε ότι εκεί καταποτούν τα άνθρωπινα δικαιώματα, αλλά κλείνουμε τα μάτια και δίνουμε λεφτά και πολλά λεφτά, ούτω ώστε αυτό το κράτος που προβέζει τα δικαιώματα θέλουμε να γίνει ο χωροφύλακας των συνόρων μας. Πάρα πολύ λογικά και συνεπεί όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η χώρα δεν έχει σύστημα ασύλου και όσοι θέλουν ε, προστασία ε, πάει και τους δίνει εκεί που διώκονται. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα για το ότι ε, τελικά πάνω απ' όλα η Ένωση θέλει να φρενάρει τις μεταναστευτικές ροές. Ενά, τι κάνουν τόσες πολιτικές ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Δύο μέτρα και δύο σταθμά και αυτά θέλουν να τα ενσωματώσουν στο ψήφισμα. Στέτινα και ολοκληρώνουμε τη λίστα των συντακτών. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ελεύθερα ΜΜΕ, ανεξάρτητος τύπος. Αυτά είναι οι εχθροί του Λουκασέγκο. Δημοσιογράφοι με ανεξάρτητα ΜΜΕ, αυτά είναι ο στόχος. Εκφοβισμός, αυτή η διαδικτυακή πύλη έχει μπλοκαριστεί τόσο καιρό και επίσης το 10 είχαμε ε, κάποιον από το χάρτη 97 που δολοφονήθηκε και τελικά αναγκάστηκαν να πάνε στο, στην Πολωνία. Βλέπετε ότι μετά ακολούθησε ένα κύμα κατασχέσεων, ερευνών ε, και ε, συναμβάνονται και φυλακίζονται οι δημοσιογράφοι, γύρω στους 100 συνελήφθησαν ε, πέρσι. Πριν από δύο χρόνια ε, ήραμε του περιοριστικά μέτρα κατά της χώρας και επομένως μπορούν να έχουν ε, ένα σωρό χρήματα από εμά χωρίς προϋποθέσεις. Μα θα έπρεπε να έχουν προϋποθέσεις ελευθερίες και δικαιώματα. Αντί να εκδημοκρατήσει τη χώρα, ο Λουκασέκο κάνει τα πράγματα αυστηρότερα διώκει αυτούς που προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο. Μα να μην εμπιστευόμαστε δικτάτορες. Αυτή η πύλη χάρτη 97 είχε αφορμή ένα κίνημα που εμπνεύστηκε από το τσεχοσλοβάκικο χάρτη 70 και ως τσέχος θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να καταπολεμήσω την καταπάτηση των δικαιωμάτων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 ως ε, πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας ε, με την Λευκορωσία δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι υπόλοιποι βουλευτές θα τονίσω ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Λευκορωσία είναι και δικαίως υπερήφανη για τους καλλιτέχνες της να έχει και ένα Νόμπελ ε, λογοτεχνίας αλλά το θέατρο στην ε, Λευκορωσία υποφέρει μιλάω για το ελεύθερο θέατρο Λευκορωσίας το οποίο καταπιέζεται με διάφορους τρόπους καλλιτέχνες, καθηγητές ε, και όσοι θέλουν να βοηθήσουν το θέατρο αυτό καταστέλλονται πρέπει λοιπόν να συντάξουμε μια γνωμοδότηση που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Ευχαριστώ. Την ομάδα των σοσιαλιστών το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τζούλι e action. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για το θέμα της ε, Λευκορωσίας. Η παθητικότητα της ε, Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έχει πλέον αποθρασύνει την κυβέρνηση Λουκασέγκο. Ειδικά η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, επιδεινώνεται και η μεταχείριση των πολιτικών αντιπάλων είναι φρικτή σε μια χώρα όπου η θανατική ποινή παραμένει. Η περίπτωση του Μιχαήλ Ζανσούσνη είναι ιδιαίτερος αποτρόπαια. Είναι στην απομόνωση από τον Ιούλιο σχεδόν στην Ευρώπη αυτά. Ο Δημήτρη Μπόμπρικ που συνελήφθη τον Αύγουστο έχει πει πως ε, ενώ ήταν κρατούμενος τον ανάγκασαν να υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας με την ΚΑΓΕΜΠΕ στην περίπτωση του Χάρτη 97, τα ακούσαμε ήδη. Και εγώ έχω συνεργαστεί με αυτή την οργάνωση τους τελευταίους μήνες και πραγματικά αισθάνομαι ότι τους έχει προδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητάω από τον Επίτροπο Χάν και την ύπατη εκπρόσωπο να αναλάβουν δράση και να απαιτήσουν βελτιώσεις στα θέματα αυτά την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος Γιούρεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Λευκορωσία είναι ένας κοντινό μας γείτονα και πολύ σημαντική χώρα. Χώρα που έχει κοινά σύνορα με πολλές Ευρωπαϊκέ. Το έθνος της Λευκορωσίας αγωνίζεται για την ιστορική του μνήμη μεταξύ άλλων βάσει του Norman Davis, ενός Βρετανού ιστοριογράφου, 250.000 ε, ε, άνθρωποι στη Λευκορωσία δολοφονήθηκαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Τώρα φαίνεται ότι αυτό ε, δεν ε, γίνεται καν σεβαστό ή γνωστό. Σταυροί δεν έχουν μπει στους τάφους των θυμάτων αυτών, διότι δεν ε, είναι γνωστό που είναι θαμένοι καν. Θα έλεγα λοιπόν στις αρχές της Λευκορωσίας να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Πάψτε την σύλληση αυτού του νεκροταφείου, διότι είναι ένα έγκλημα που μας ενοχλεί όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση του τύπου στη Λευκορωσία διαρκώς επιδεινώνεται. Η Λευκορωσία αυτή τη στιγμή είναι 155η από τις 180 χώρες ε, για την ε, ελευθερία της δημοσιογραφίας. Οι συλλήψεις, οι εκφοβισμοί, οι απειλές είναι μέρος της καθημερινότητας των εξάρτητων δημοσιογράφων στη χώρα. Στις αρχές του Αυγούστου του 2018 οι αρχές της Λευκορωσίας ε, πραγματοποίησαν επιδρομή στον ανεξάρτητο σταθμό τις χώρες Μπέλτα ε, και υποχρέωσαν όλοι να ε, γραφούν σε κατάλογο για να χάσουν την ανωνυμία τους προτού μπορέσουν να έχουν άδεια λειτουργία. Αυτό αντίκειται σε όλες τις αρχές που περασπίζονται όλοι σε αυτή την αίθουσα. Επίσης, ε, ήρθε η απαγόρευση της που χάρτης 97. Ζητώ λοιπόν να ε, συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις με οργανώσεις στη Λευκορωσία γιατί το χρωστάμε στους πολίτες της χώρας. Πρέπει να προασπιστούμε την ελευθερία της έκφρασής τους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό για την ομάδα της αριστεράς η κυρία Βερζιά. Για 1,5 λεπτό, συγγνώμη κυρία Βερζιά, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η η Λευκορωσία θεωρείται ως η τελευταία δικτατορία της Ευρώπης, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η θανατική ποινή ισχύει. Δεν υπήρξαν εκλογές που να ε, συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα από το 2001. Ο κ. Λουκασένκο επανελέχθη το 2015 με 83,5% των ψήφων. Ναι, λοιπόν, καταπιέζονται τα... Ε, τα παραδείγματα καταπίεσης του τύπου, μεταξύ των οποίων και ο χάρτης 97. Το καθεστώ απελευθέρωση των θεωρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δείγμα αφέλεια. Όχι. Είναι ίσω υποκρύπτει κάποια συμφέροντα. σω. σω όμω να είναι χωροφύλακα τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Λευκορώσια. Τα εργαλεία γειτονία και τα κονδύλια του έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο των σύνορων και όχι σε άνοιγμα. Και αυτό βεβαίω ε, ε, είναι κάτι που και η πολωνική κυβέρνηση επιδιώκει. Οι Τσετσενοί, οι Σύριοι και άλλοι που φτάνουν στη Λευκορωσία περνούν από εκεί τα σύνορα. Οι Πόλωνοι έχουν αρνηθεί τι αιτήσει ασύλου και πολλοί έχουν ε, αναπευθεί προ τη Ρωσία ιδίω. Ε, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα για τους Ουκρανούς εργαζομένους που έχουν άδειε ε, παραμονής από τον Νότο ε, για να εργαστούν αλλά δεν βλέπουν την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη πέρα από τα σύνορα αυτής της χώρας. Θα πρέπει επαναπρόθεση σε χώρες όπου καταγγέλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να πάψει. Να πάψει. Η ανακολουθία μας, δύο μέτρα και δύο σταθμά, πρέπει επίσης να σταματήσει και να σταματήσουν να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ορισμένων κατώμελων. Και ο κύκλος εκ μέρους των πολιτικών ομάδων το λόγο έχει η κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, η κοινωνία ε, έχει όση ελευθερία έχουν τα μέσα ενημέρωσής της. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τα ελεύθερα ΜΜΕ. Τώρα όμως στη χώρα υπάρχει καινούριο κύμα καταστολής και όποιος αντιπολιτεύεται τον Λουκασέγκο πάει φυλακή, ε, ξυλοκοπείται, υφίσταται χρηματικές ποινές. Ναι, αυτό έγινε και με τον Χάρτη 97, αυτή την πλατφόρμα για τη δημοκρατία στη χώρα. Τον Ιούνιο φέτος το Κοινοβούλιο ενέκρινε ε, νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωση. Ε, αυτός ο νόμος υπό το ένδυμα της καταστολής των ψευδών ειδήσεων αποτελούσε θεσμοποίηση και θεσμοθέτηση της λογοκρισίας. Θα πρέπει αυτές οι ελευθερίες να είναι προϋπόθεση της συνεργασίας μας. Intimidatie, arrestaties εκφοβισμός, ε, συλλήψεις, ε, λογοκρισία. Όλα αυτά έχουν φέρει την Λευκορωσία στην 155η θέση στον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου. Ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη, ο Λουκασένκο, κυβερνά 24 χρόνια ήδη. Έτσι είχαμε και τις ειρηνικές διαδηλώσεις ε, του Φεβρουαρίου του 2017, οι οποίες καταστάλησαν 700 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 100 δημοσιογράφοι. Και συνεχίζεται ακόμα ο εκφοβισμός των ΜΜΕ. Ας μην είμαστε λοιπόν αφελείς. Ο Λουκασέγκο δεν ενδιαφέρεται για μεταρρυθμίσεις. Θέλει μόνο περισσότερα λεφτά, περισσότερη εξουσία και αναγνώριση. Αυτό κάνει μόνο καταλαβαίνει λοιπόν μόνο ξεκάθαρη γλώσσα. Όσο δεν σέβεται την ευθεία του τύπου δεν μπορούμε να μιλάμε για προσέγγιση. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί τέσσερα αιτήματα. Τα κάνω και τα τέσσερα αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Φαρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ θέλω να μιλήσω για την ε, καταπίεση συγκεκριμένη ε, δηλώτριας από την περασμένη χρονιά που είχε εκφραστεί κατά του δικτάτορα Λουκασένκο. Οι δικαστικές διώξεις, η καταπίεση των ε, blogger και των ελεύθερων δημοσιογράφων είναι πραγματικά η καταπίεση της ελευθερίας, ε, των δημοκρατικών αξιών και όσων προασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέφουμε στον τρόπο λειτουργία και την απολυταρχία των προηγούμενων καθεστώτων. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για το μόνο καθεστώς στην Ευρώπη που ακόμα εφαρμόζει τη θενατική ποινή και έχει και τα σχέδια για την οικοδόμηση του πολιτικού σταθμού στο Όστραβετς. Θα πρέπει λοιπόν να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας με τη Λευκορωσία μόνον εφόσον γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2004 είχαν λάβει το βραβείο Ζαχάροφ ε, η ομάδα των Λευκορώσων δημοσιογράφων. Θα πρέπει λοιπόν τώρα κατηγορηματικά να καταδικάσουμε όλες αυτές τις ε, παραβιάσεις ελευθεριών τους. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Πόλτσακ. Ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να καταδικάσω τα όσα κάνει η κυβέρνηση Λουκασέγκο που καταπιέζει την ελευθερία τύπου και έκφρασης Μερικές φορές ε, κοιτάμε κάποια πράγματα και ξεχνάμε ότι μιλάμε για διαφορετικούς πολιτισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι γίνεται στην ε, γειτονιά μας χωρίς να θέλω να μειώσω την ε, σημασία των πιο απομακρυσμένων περιπτώσεων παραβίασης. Οπωσδήποτε η ελευθερία του τύπου είναι μια δημοκρατική αξία και θα ήθελα να την στήριξω και με την ψήφο μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρω. Εάν είναι να γίνουμε καρφιά στο φέρετρο του τυράννου ευχαρίστως να γίνω. Αυτά είναι τα λόγια του Όλαξένσο Ουκρανού σκηνοθέτη που βρίσκεται στην Ουκρανία αλλά ισχύουν και για το χάρτη 97 και άλλους ανεξάρτητους μουσιογράφους έχουν γίνει τα καρφιά στο φέρετρο του πολιτικού κατεστημένου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μια συμφωνία καλής βούλησης και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στις αρχές της χώρας τις υποσχέσεις τους για τα ζητήματα αυτά. Ένα σημάδι θετικών εξελίξεων θα είναι το ξεμπλοκάρισμα του χάρτη 97 και να σταματήσει ο εκφοβισμός των ανεξάρτητων ΜΜΕ και να αποσυρθούν οι ψεύτικες κατηγορίες. Αν δεν γίνουν σεβαστές αυτές οι δεσμεύσεις, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει αποφασιστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. κύριος Ιτουργκάης Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για μια δικτατορία του 21ου αιώνα στην Ευρώπη και ακριβώς έχουμε εκεί πέρα καταστολή, έχουμε απειλές κατά όποιου παλεύει για την ελευθερία και τα δικαιώματα, αλλά επίσης έχουμε καταστολή και απειλές για τα μέσα ενημέρωσης που θέλουν ελεύθερα να ενημερώνουν για τα όσα γίνονται σε αυτή την ευρωπαϊκή χώρα. Λένε ότι ο Θεός τους πλάθηκε ότι ομοίως Αϊ πελάζει. Να, και με, είναι φίλος του του Λουκασέγκο ο Μαδούρο. Που τα ίδια κάνει και αυτό στη Βενεζουέλα. Να, είδατε τι είναι με το Χάρτεν 97. Θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Ε, πέρασαν κάθε κόκκινη γραμμή. Και οι προς την κυβέρνηση αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα να κλείσει η κυρία Μπιενκόφσκα. Σας ευχαριστώ. Οι σχέσεις ε, των δύο μερών ε, θα πρέπει να συνεχίσουν με την βάση της ε, επαφής με κριτική που ασκούμε. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η πρόοδος σε διάφορους τομεί ε, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Λευκορωσίας έχουν προχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συμμετοχή τη Λευκορωσίας στην Ανατολική Γειτονία και βλέπουμε ακριβώ επανάληψη του τομεακού διαλόγου τη εταιρική σχέση κινητικότητας των διαπροσωπικών επαφών ε, με τις ανταλλαγές όπως το Erasmus Plus, ορίζοντας 2020 ε, κτλ. Και τώρα κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε το έγγραφο κοινών προτεραιοτήτων, ένα σημαντικό κομμάτι των ε, σχέσεών μας και βεβαίως εδώ πέρα παίζουν σημαντικό ρόλο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε δει ότι οι αρχές της χώρας θέλουν να εμπλακούν επικοδομητικά σε έναν διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το είδαμε αυτό και στην τελευταία μας συνάντηση στις 17 Ιουλίου στο Μίνσκ. Στηρίζουμε επίσης την εμπλοκή για τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Η ταμενία της αυτού του διαλόγου καλύπτει επίσης τις ανησυχίες για τους ε, δημοσιογράφους ε, στην Λευκορωσία και την έλλειψη νομοθεσίας για αυτό το θέμα. Και ακριβώς θα πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά της ελευθερίας των ΜΜΕ. Θα πρέπει ακριβώς να επαναλάβουμε άλλη μια φορά τη σημασία της ελευθερίας έκφρασης και της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ. Ζητάμε ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γνωρίζουμε ότι πολλά ανεξάρτητα ΜΜΕ εργάζονται σκληρά για να επιτύχουν σοβαρά αποτελέσματα στην προστασία των δημοκρατικών αξιών και εκτιμούμε το έργο τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει στις αρχές της Λευκορωσίας πως η καταστολή των ανεξάρτητων ΜΜΕ όπως του χάρτη 97 είναι αντίθετη με τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ένα μορατόριο στην θανατική ποινή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. θα συνεχίσουμε λοιπόν την πολιτική επαφών και θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην χώρα και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Λευκορωσία στον τομέα του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά την κοινωνία των πολιτών μέσω των σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλίων. Τα βήματα που κάνει η Λευκορωσία για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα διαμορφώσουν την αντίδρασή μας. Να προσθέσω κάτι ακόμα, καθώς σήμερα συζητάμε μετά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η πυρηνική ασφάλεια είναι σημαντική. Εμείς συζητάμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για την οικοδόμηση του ποινικού εργοστασίου στο Στρόβιετ και χρηματοδοτούμε ειδικού που βοηθούν ε, τους νέους εθνικούς κανόνες για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Έχουμε λάβει έξι ε, σχέδια ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει αργότερα σήμερα. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ιδίω η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αχμέντ Μανσούρ. Ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο είναι η κυρία Λόχ Μπίλερ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω περιμένετε κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα στην οθόνη ναι ευχαριστώ εγώ θα ήθελα να μιλήσω στα κατεπήγοντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τώρα έχει διορθωθεί λοιπόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραβιάζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα συλλαμβάνονται οι επικριτές της κυβέρνησης και σύμφωνα με την ε, Διεθνή Αμνηστία ε, τα άτομα κρατούνται υπό συνθήκες ε, που ουσιαστικά αγγίζουν τα όρια του βασανισμού. Τον Μάιο ο Αχμέντ Μανσούρ καταδικάστηκε στο Αμπουντάβι σε ποινή φυλάξης δεκαετών και κατηγορούνταν για πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι η ελεύθερη έκφραση γνώμης ο Αχμέτ ε, Μανσούρ βεβαίως υφίσταται διώξεις εδώ και χρόνια και οι ειδικοί από την φυλάκισή του το Μάρτιο του 2017 ζητούν την άμεση αποφυλάκισή του. Μαζί του κρατούνται και άλλοι μη βίαιοι αντιφρονούντες. Ζητάμε λοιπόν την άμεση απελευθέρωση του Αχμέτ Μανσούρ όπως επίσης και των άλλων μη βίαιων αντιφρονούντων. Είναι πολύ περίεργο το ECR και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μην στηρίζουν αυτό το ψήφισμα. Απευθύνω λοιπόν έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να κινητοποιηθούν για την απελευθέρωση του Αχμέντ Μανσούρ και να υπερψηφίσουν το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστούμε. Έχετε δίκιο. Εγώ έκανα λάθος. Μιλούμε για τα ΙΑΕ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ιδίως στην περίπτωση του Αχμέντ Μανσούρ. Η οθόνη μου δείχνει κάτι διαφορετικό και μπερδεύτηκα. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπασίρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δώστε προσοχή σε αυτό που λέω λοιπόν και όχι σε αυτό που γράφει η οθόνη. Κύριε Μπασι, Πρόεδρε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι βασικό σύμμαχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον Αραβικό κόλπο. Πρέπει όμω να θυμόμαστε ότι όταν τα ΙΑΕ έκοψε του δεσμού από εμά ε, πέρσι. Ο Γενικό Εισαγγελέα τη χώρα προειδοποίησε ότι οι πολίτε που εκφράζουν συμπάθεια προ το Κατάρ, α πούμε, θα ε, αντιμετωπίσουν πρόστιμα και ποινή φυλάκιση ω 15 χρόνια. Υπ' αυτήν την έννοια, η ολομέλειά μα πρέπει να είναι απολύτω ξεκάθαρη. Η ελευθερία έκφραση και ο σεβασμό των ελευθεριών των πολιτών δεν είναι απλώ θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει να κάνει με την ε, προστασία της ειρήνης και της ευμερίας της όλης περιοχής. Το κάτας δικαίου έχει σημασία για την προστασία των πολιτών από τις αδικίες της κυβέρνησης και του κράτους. Και όχι αντιστρόφως, μπορώ λοιπόν να πω ότι μόνο εάν τα ε, ε, συμμορφωθούν με τις δηλώσεις του ΟΗΕ για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους επιτρέπουν να δρουν, τότε μόνο μπορούμε να τους ξαναδούμε στο ΝΟΙΑ για να προωθούμε την ειρήνη, την ευημερία και την ε, σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε και Ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο ομιλία σα. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Πόστ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε καιρού που βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμό των ε, ακτιβιστών ε, που πέφτουν θύματα επειδή κάνουν απλώ τη δουλειά του, δεν εκπλησόμαστε. Ανησυχούμε όμω πάρα πολύ για όσα συμβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Αχμέτ Μαζούρ βρίσκεται στη φυλακή γιατί υποτίθεται ότι δημοσίευσε ψευδείς πληροφορίες για να καταστρέψει την ε, καλή φήμη των ΙΑΕ στο εξωτερικό. Όμω αυτό που πραγματικά καταστρέφει τη φήμη του των ΙΑΕ ε, στο εξωτερικό είναι το πώ φημώνουν την ελευθερία τη έκφραση. Ζητούμε την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση του Αχμετ Μαζούλ και όλων των άλλων ακτιβιστών και αντιφρονούντων. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουν να εμπορεύονται όπλα και εξοπλισμούς ασφάλειας με τα ΙΑΕ. Πώς μπορούμε να διατηρούμε το πρόγραμμα ε, διευκόλυνσης των θεωρήσεων με την χώρα αυτή όταν είναι σαφές ότι παραβιάζουν τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι μέρος της συμφωνίας. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει την ε, την συμπεριφορά προς τον Μανσούρ και να καλέσει στην άμεση απελευθέρωσή του. Το ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, έχει ως πρώτη στη αξία τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εμπορικές και διεθνείς μας συμφωνίες. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Σχάκε. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι φιλοδοξίες των Αραβικών Εμμυράτων μοιάζουν ατελείωτες. Λένε ότι είναι μια χώρα νεανική με υψηλή τεχνολογία που έχει επιτύχει εκπληκτική ανάπτυξη, αναζητεί πιο ενεργό ρόλο. Έχει όμως μεγάλη σημασία η φήμη των Αραβικών Εμμυράτων και είμαι πεπισμένη ότι η σύλληψη του Αχμέντ Μασούρ για κάποια tweet και η αντιμετώπιση του δεν έχουν βοηθήσει ως προς αυτό. Αλλά βεβαίως ε, στόχο μας δεν είναι να δώσουμε στην χώρα αυτή συμβουλέ δημοσίων σχέσεων. Ο κύριο Μανσούρ έχει αναγνωριστεί ως ένας θαραλέο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κέρδισε το βραβείο Μάρτιν Άναλ και ήταν σύμβουλο του Human Rights Watch. Τώρα είναι στην απομόνωση. Και δεν μπορεί να ε, έρθει σε επαφή με κανέναν. Δεν έχει καν δικηγόρο και έχει ανακληθεί και το διαβατήριό του. Γύρω στο 1 εκατομμύριο δολάρια έχουν επενδυθεί σε ένα Ισραηλινό σύστημα παρακολούθησης των επικοινωνιών του κυρίου Μανσούρ. Θεωρώ ότι τέτοια συστήματα που φτιάχνονται και στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να εξάγονται σε χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι κάνουμε με τις εξαγωγές στην περίπτωση του κυρίου Μανσούρ. Βλέπουμε, θεωρούμε ότι οι δράσεις του είναι απλά έκφραση γνώμης και ζητάμε από τις αρχές της χώρας να τον απελευθερώσουν. Επίσης, θα πρέπει να επανεξεταστεί ο νόμος περί κυβερνοεγκλήματος για να συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές. Επίσης, η κυρία Μογκερίνη θα πρέπει να μιλήσει με λόγια σταράτα για την περίπτωση Μανσούρ και για όσους σκοπεύουν να πάνε διακοπές στα Εμμυράτα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν το τι συμβαίνει αφού στείλουν ένα tweet που θα ζητάει εκλογές. Δεν μου φαίνεται και πολύ φιλόξενη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βερζιά για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ και πολύ καιρό δεν έχουμε βάλει σημείο στη διάταξη το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα. Γιατί είναι η μόνη χώρα στη χώρα που έχει τύχη απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατήριων. Ε, εκεί δέχονται ε, πάρα πολλού μετανάστε, 5% στο Ντουμπάι και είναι πάρα πολλοί δυτικοί που δουλεύουν εκεί σε πολυεθνικέ. Βέβαια παρά τα διπλώματα υπάρχει θεσμένη ε, διάκριση, περισσότεροι είναι εργάτε τους ε, προσλαμβάνουν για τα φρονικά έργα και είναι θύματα κυρίως οι γυναίκες αυτής της ε, μοντέρνας δουλείας. Τα Μοιράτα είναι καλοί πελάτες Το Ισραήλ και η Γαλλία τους δίνουν ε, τεχνολογία για να κατασκοπεύουν. Και το ίδιο ισχύει και για τους ακτιβιστές των ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, βέβαια όπλα τους δίνει κυρίως η Γαλλία και υπάρχει πάρα πολύ διαφθορά που ξεσκέπασαν τα ΜΜΕ της Γαλλίας. Ε, αυτά χρησιμοποίησαν στην Ιεμένη ε, και υπάρχει λάθρο εμπόνιριο και μες στην ανθρωπιστική κρίση εμπάργο στα όπλα και να πετηθεί να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους και να αποφυλαγήσουν τους ακτιβιστές. ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ΕΛΚΑΝΕΚΑΔΕΝ ήταν με το μέρος των καταπιεσμένων για όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο. Οπότε ξέρουμε τι συμβαίνει με τον Μανσούρ, είναι να τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταδικάστηκε σε κάθερξη για παραπληροφόρηση, διατάρξη της ειρήνης, για όλα αυτά τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν εγκλήματα. Κάθερξη, 10 χρόνια μέσα. Και συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να τους βάλουμε κάτω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τους πούμε ότι παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Το ΕΛΚ δεν είναι ικανοποιημένο από το τελικό κείμενο. Και αντί να αναφέρουμε γεγονότα, ε, το κείμενο είναι γεμάτο με χαζομάρες ε, ιδεολογικές και σε πέντε λεπτά όλα αυτά μπορεί να τα γκρεμίσει κανείς έτσι με το Google. Θα πρέπει να έχει πιο πολύ αξιοπιστία το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε στα ψηφίσματά μας να στηριχθούμε σε πραγματικά περιστατικά και όχι ιδεολογήματα. Κύριε Στεχόφσκι, μίλησατε και ω Συντάκτη και ω ΕΛΚ. Και τώρα η κυρία Γουόρντ για ένα μισή λεπτό. Συνεχίζει να επιδεινώνεται η κατάσταση στον ε, κόλπο. Τα κράτη με τα θα πρέπει αποφασιστικά να ανασχέσουν αυτές τις κατα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί πρόκειται για κράτη εταίρους μας και είδατε τι έγινε με τον κύριο Μανσούρ, τα είπαμε στην αρχή του έτους, ε, Φοβόμαστε και τελικά δικαιώθηκαν οι φόβοι μα για αυτή την ε, κακομεταχείριση που υφίστατο ενώ ήταν στη φυλακή. Συνηθισμένα πράγματα. Είχαμε πληροφορίες ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την οικογένεια, με του συνηγόρου του και τα Εμμυράτα θα πρέπει άμεσα και χωρίς όρους και προϋποθέσεις να τον αποφυλακίσουν, να ε, καταπέσουν όλες οι κατηγορίες. Απλώς εξέφρασε απόψεις στα κοινωνικά μέσα. Να σταματήσουν επίσης και οι δυσμενείς διακρίσεις κατά των γυναικών εκεί. Περιστέλλεται η ελευθερία τους και ακόμα α, τελούν υπό την επιτροπή των ανδρών καταστολή, επιθέσεις και παρεμπόδιση των ακτιβιστών των δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα εργασιακά δικαιώματα και έχουμε συνεχώς παραβίαση του εργατικού δικαίου από τους εργοδότες. Θα πρέπει να τους πούμε ότι πρέπει να τα πάνε καλύτερα σε αυτό το μέτωπο γιατί εκεί επενδύουμε δισεκατομμύρια άρα έχουμε ευθύνη Πρέπει να απαιτήσουμε να βρουν ε, εκεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενάμιση λεπτό ο Σουρμπάν Κρέσπο. Το 15 ο Μανσούρ κατήγγειλε ότι στη χώρα φυλακίζονται όσοι είναι αντιπολίτευση. Σεξουαλική βία, βασανιστήρια, να αποσπάσουν ομολογίες καταδίκες χωρίς δίκη. Και τώρα για ε, δημοσιεύσεις πάλι έχουμε φυλακίσεις και βασανισμούς. Μιλάμε για παραβίαση δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος. Εκεί ε, με την πρόφαση καταβλήμησης τρομοκρατίας και τα πιο βασικά δικαιώματα δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Και εκεί αυτό το οποίο κάνουν είναι να χρησιμοποιούν όπλα και τεχνολογία κατασκοπίας που τους έδωσε η Ευρώπη, ούτω ώστε να μπορούν να ασκήσουν αυτή την καταστολή. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούσαν να καταστήλουν το λαό. Τον ίδιο το Μανσούρ τον κατασκόπευαν με τέτοιο λογισμικό. Οπότε τελικά έχουμε και απελπισία και ο εξτρεμισμός έτσι γεννάται. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να προκαλούμε έμεσα αυτήν την απελπισία. Να σταματήσουν τα βασανιστήρια. Να κάνουμε εμπάργο και για τα όπλα και για αυτό το λογισμικό κατασκοπίας. Να σταματήσουμε να είμαστε συνένοχοι στα Εμμυράτα τέρμα στις δηλώσεις. Να εφαρμόσουμε εμπάργκο στα όπλα. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ όμως να είστε πιο πειθαρχημένοι επόμενοι σε ό,τι αφορά το χρόνο αγόρευσης. Κοράω για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και η τελευταία ελεύθερη φωνή των Αραβικών Εμμυράτων ε, σιώπησε. Ο Αχμέτ Μανσούρ ήταν ο τελευταίο ακτιβιστή που είχε μείνει στα Εμμυράτα και που τολμούσε δημόσια να αμφισβητήσει τι αρχέ. Και αυτό το πλήρωσε με καταδίκη δεκαετού ε, κάθερξη. Μπορούμε ακόμα να ανεχόμαστε αυτή τη στάση των Αραβικών Εμμυράτων απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και από την άλλη πλευρά, τι μπορούμε να περιμένουμε από μια χώρα που τοποθετείται στο 100, 100 ε, στη 16η θέση στο, στο δίκτυ παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα που είναι πρωταθλητής για την παγκαταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τον αντιτρομοκρατικό νόμο που περιλαμβάνει μια έναν ευρύτατο ορισμό του αδικήματος αυτού, ώστε να, μπορεί, να μπορούν οι αρχές να διώκουν οποιοδήποτε θέλουν ε, και τους ε, ακτιβιστές και όποιους άλλους αντιφρονούνται. Συστηματικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό ο νόμος για να ελέγχονται οι πολιτικοί αντιφρονούντες. Η Κομισιόν θα πρέπει να ε, προβεί σε αίτημα για την άμεση απελευθέρωση του Μανσούρ και άνεφόρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ζαν Λουκ Σαφχάουζεν, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένε από τι χώρε μα έχουν καταλάβει πόσο θανάσιμος κίνδυνο είναι τα Εμμυράτα με άλλες χώρες που ε, έχουν ορίσει την οργάνωση του Μανζούρ ω τρομοκρατική. Ενώ είναι διπλή η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αυτοί δείχνουν διάβια και προστατεύουν τους πληθυσμούς τους. Χειρίζονται... <coughs> Υπάρχει βέβαια χειρισμός από πλευράς του Κατάρ που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένους ε, ε, ε, τη συγκεκριμένη οργάνωση. Ο κύριος Μανσούρ είναι συνδεδεμένος με τους αδερφούς μουσουλμάνους. Goal for Human Rights επίσης συμμετέχει εκεί, χρηματοδοτείται από τον κύριο Σόρο ε, που χρησιμοποιεί τα χρήματά του για να στηρίξει τρομοκράτες ώστε να βλάψει τα δικά μας κράτη. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Προσθέτω ότι πρόκειται για έναν που επανελειμμένος έχει ε, προβεί σε τέτοιου είδους ε, πράξεις. Ευχαριστώ. Καν. Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε με Μανσούρ έχει γίνει σύμβολο της καταστολής της ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεστε στα Ηνωμένα Αραβικά Έμυρα. Το παρενοχλούν, τον διώκουν εδώ και χρόνια πριν την πρώτη του σύλληψη το 2011, οπότε είχε ζητήσει πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Τον Μάιο καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθερξη επειδή εξέφρασε απόψεις του στο Twitter. Προσπαθούν τα Εμμυράτα να παρουσιάζουν μια εικόνα ανοίγματο και σύγχρονου κράτου. Ε, Παρακαλώ λίγο πιο αργά να μιλάτε, λέει ο Πρόεδρος. Λίγο πιο αργά να μιλάτε, παρακαλώ. Υπάρχουν φωνές αντιφρονούντων που δεν επιτρέπεται να ακουστούν ε, χωρίς να φοβούνται αντίπεινα. Το στην περιοδική ε, αναθεώρησή του, ο ειδικό απεσταλμένος έκανε πολύ αρνητικές κριτικές. Ζητούμε άμεση απελευθέρωση του Μανσούρ. Σύμφωνα ε, με το Διεθνές Δίκαιο δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο από ένα κράτος που είναι μέλος ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγγίλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ήδη έχουμε ακούσει για τον υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αχμέτα Μανσούρ που έχει μπει στη φυλακή για 10 χρόνια επειδή άσκησε το δικαίωμα τη ελευθερία έκφραση online. Το έγκλημά του ήταν να προωθεί στην ελευθερία έκφραση, στην ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών στη χώρα του και όχι απλά αντιμετώπισε σημαντικέ και επανειλημμένε απειλές σα και τα κτλ. αλλά περιορίστηκαν και ανεστάλησαν τα πολιτικά του τα αφρικά δικαιώματα. Ε, τιμωρήθηκε τελικά ε, και μπήκε και φυλακή. Βλέπουμε ότι τα σώματα της ασφάλειας ε, στη χώρα στοχεύουν τους ακτιβιστές και τους περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε απαγωγές από αρχές ασφαλείας ε, που δεν δίνουν σε κανέναν λογαριασμό για τις πράξεις τους. Ερώτηση προς την Κομισιόν, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει ε, τέτοιους αγνοούμενους ε, όταν συζήτησε συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά επίσης. Έχει κάνει έκκληση στον το δικαστήριο όμως απέναντι στην ποινή. Πώς θα εξασφαλίσουμε μια δίκαιη δίκη. Τέλος, ε, η ε, νομοθεσία για την ε, αντιμετώπιση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που εγκρίθηκε ε, εισάγει ακόμα πιο αυστηρές ποινές και κυρώσεις. Ηλεκτρονική επιτήρηση ακτιβιστών είναι... διακόπτεται η ομιλήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θέλω να ζητήσω από τους ομιλητές να πειθαρχούν στο χρόνο τους. Περνάμε στη διαδικασία Catch ε, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ο Αχμέντ Μανσούρ είναι μία από τις τελευταίες φωνές που ανοιχτά επικρίνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά από απειλές θανάτου, αυθαίρετα συλλήφθηκε και καταδικάστηκε σε 10 έτη φυλάκισης. Το έγκλημα αυτού του ακτιβιστή είναι ότι ειρηνικά διεκδικούσε στα, στα κοινωνικά δίκτυα ε, και αγωνιζόταν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αφήσει, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, να φυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός και οι υπόλοιποι αντιρρησίες συνείδησης ή αντιφρονούντες σε αυτά τα ε, καθεστώτα. Θα πρέπει να καταργηθούν τα βασανιστήρια και η θανατική ποινή και να ε, γίνουν σεβαστές οι ατομικές ελευθερίες αλλά και η ελευθερία έκφρασης πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριο Ευχαριστώ πολύ Υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την οικονομία κτλ. Όμως, συγχρόνως, δεν υπάρχει ελευθερία για όλους στη χώρα. Και αυτό είναι το αρνητικό. Και αυτό ισχύει και για τον Αχμέτ Μανσούρ. Είναι κρατούμενος γιατί θέλει να εκφράσει τις απόψεις του στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν συμφωνεί η κυβέρνηση, δεν της αρέσουν τα σχόλια και τώρα βρίσκεται στη φυλακή για πολύ καιρό. Και δεν ξέρει πότε θα απελευθερωθεί. Καλό είναι που συζητάμε για αυτή την υπόθεση σήμερα το πρωί εδώ και πρέπει να πιέσουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να τον ελευθερώσουν. Έχουν πετύχει μεγάλη πρόοδο στην οικονομία τους αλλά οι βασικές ελευθερίες θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Επόμενος, ο κύριος Μαριάς. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Αραβικής Κερσονήσου, δεν υπάρχει κάνει έννοια της δημοκρατίας διότι εκεί υπάρχει πλήρης καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι ακτιβιστές βασανίζονται οι bloggers διώκονται υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τους αντιφρονούντες όλα αυτά βεβαίως για τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα όπου συνεχίζονται οι διακρίσεις κατά των γυναικών και φυσικά δεν τηρούνται οποιαδήποτε εργασιακά δικαιώματα. συνεχίζει να υπάρχει η θανατική ποινή νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να στείλει ένα αποφασιστικό μήνυμα η ευρωπαϊκή ένωση προς τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα τα οποία συμμετέχουν στη σφαγή που γίνεται στην ιεμένη στα οποία αραβικά εμιράτα πωλούν όπλα οι ευρωπαϊκές εταιρείε πώλησης όπλων και παραγωγής όπλων. νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προ τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα όχι χαϊδέματα πλέον προ αυτού από την ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Καστάλντο. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, επιτέλους καταφέρνουμε να μιλήσουμε για τον Αχμέτ Μανσούρ, blogger από τα Εμμυράτα, που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν τελευταία ανεξάρτητη φωνή που δεν είχε φυλακιστεί και κατήγγειλε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Εμμυράτα. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση επειδή δημοσίευσε στα κοινωνικά μέσα ε, λάθος ψευδείς πληροφορίες ε, ε, ε για μίσους. Ε, κατά τη γνώμη μας ειρηνικά προσπαθούσε να αντισταθεί. Αλλά αυτό που ακόμα περισσότερο εντυπωσιάζει είναι η δική μα στάση ω Ένωση που είμαστε αμφίσιμοι και υποκριτικοί. Από τη μια πλευρά κάνουμε του πρωταθλητέ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την άλλη ε, δίνουμε και πουλάμε software κατασκοπικό σε καθεστώτα τελείως ε, αντιδημοκρατικά. Ζητάμε λοιπόν άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση του Μανσούρ και όλων των άλλων ε, αντιφρονούντων θα πρέπει σαφώς να μιλάμε όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, να σταματήσουμε την εξαγωγή τεχνολογίας, ε, κατασκοπίας και όπλων ε, προς τις χώρες αυτές. Δεν μπορούμε να είμαστε προνομιακοί συνένοχοι ε, τέτοιων καθεστώτων εις βάρος των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω λέει ο κύριο Πόλτσακ, να μιλήσω υπέρ του Αχμέτ Μανσόρ και τη απελευθέρωσή του. Αλλά θέλω να αντιδράσω και σε αυτά που άκουσα πριν. κάποιο είπε ότι καλώ μένει στη φυλακή ο κύριο Μανσούρ. Μα νομίζω ότι δεν μπορεί ένας ευρωβουλευτής να μιλάει έτσι. Εγώ το βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητικό. Για μένα είναι σημαντικό να πούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται στις χώρες του κόλπου όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορεί να σιωπούμε όταν πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κύριος Μανσόρ βρίσκεται στη φυλακή, βασανίζεται, δεν έχει δικαίωμα σε δικηγόρο. Όλα αυτά πρέπει να τα καταγγείλουμε. Βέβαια, δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με όλη τη διατύπωση, αλλά σαφώς και θέλω την απελευθέρωσή του. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρούμπικ τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για μένα διαπιστώνεται ότι η ελευθερία έκφρασης ε, ε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε όμως ε, για την ευστηκλοφορία των ανθρώπων, για τον Brexit και νομίζω ότι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχουν πολιτικοί, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και βλέπουμε ότι στην πολιτική υπάρχουν πολλοί που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και την εκτιμούν την Ευρώπη ακριβώς για το ότι προσφέρει αυτή την ελευθερία. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να κάνουμε επισκέψεις στη χώρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και εδώ στην αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επαναλαμβάνουμε συνεχώς ε, την ε, ανάγκη για να υπάρχει ελευθερία έκφραση ε, και όλα αυτά σίγουρα προάγουν και την, τον πολιτισμό και από τις εμπειρίες μου έχω ε, διαπιστώσει ότι μόνο με το διάλογο λύνονται. Ε, ή τέλο πάντων ο καλύτερος τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι ο διάλογος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Επίτροπος τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν η πρώτη χώρα με την οποία ξεκίνησε συνολικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση με 8 συναντήσεις που έγιναν ε, ήδη με τελευταίο τον Ιούλιο στο Αμπουντάμπι. Από την αρχή αρχίσαμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και βλέπουμε κάποια βελτίωση σε θέματα ισότητας, για παράδειγμα, ή θρησκευτικής ανοχής. Βέβαια, υπάρχουν ανησυχίες για πολλούς τομείς. Η θρησκευτική ανοχης βεβαια υπαρχουν ανησυχιες για έκφρασης, ε, του συνέρχεστε, οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται πολλές φορές. Αυτά είναι από τα θέματα τα οποία επανειλημμένα γύρουμε κάθε φορά που είμαστε σε διάλογο μαζί τους. Θέλουμε από αυτούς να ε, υπάρχει διαφάνεια για να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί τις δεσμεύσεις που ίδια έχει αναλάβει απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών. Παρά τις ε, αλλαγές δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αντιπροσωπεία μας ε, στο Αμπουτάμπι Παρακολουθούμε συνολικά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και βέβαια με μονομένες περιπτώσεις. Η περίπτωση του Αχμέτ Μανσούρ είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που παρακολουθούμε από κοντά. Ο κύριος Μανσούρ ο οποίος το 2015 βραβεύτηκε ως ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μάιο που μας πέρασε καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση ε, κατηγορούμενος για τα όσα εξέφρασε στα μέσα δικτύωσης και στα tweet του. Χρειάζονται διευκρινήσεις από τις αρχές των ε, Αραβικών Εμμυράτων όσον αφορά την κατάστασή του, την υγεία του, πότε θα γίνει ε, η έφεση κλπ. Έχουμε επαναλάβει ξανά και ξανά ότι η θέση μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης είναι σαφής και υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές γι' αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι θα ασχοληθούμε παρατέρω με την μεμονωμένη αυτή περίπτωση και θα εξακολουθούμε να γύρουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε φορά που έχουμε διάλογο με την περιοχή. Υπάρχουν ζητήματα και σταθερότητας που προβάλλει η χώρα, αλλά εμεί είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να υπάρχει σταθερότητα χωρί παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη θεμελιωδών ελευθεριών. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε. Έχω ψηφίσματα τα οποία θα ψηφιστούν στο τέλος της συζήτησης. Έληξε συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ψηφίσουμε σε μισή ώρα περίπου. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το επόμενο κατεπήγον, που είναι οι μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάκων στην αυτόνομη περιοχή Σιντσιάνγκ των Ουιγούρων. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μπουτικόφερ. 1,5 λεπτό. Ο συντάκτης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η κομμουνιστική ηγεσία της Κίνας στο Γιάνγκ έχει δημιουργήσει ένα αστυνομικό κράτος, ε, εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω πάνω από ένα εκατομμύριο ε, Κινέζοι ε, πολίτες που κατάγονται, έχουν η καζική καταγωγή, κατοικούν. Και λένε ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Κανείς μπορεί, ναι, να την αντιμετωπίσει τρομοκρατία με πλήρη καταστολή τουλάχιστον να υπάρχει αρκετό ε, νερό για να μπορούν να ε, κολυμπούν σαν ψάρια οι τρομοκράτες. Όχι. Αν θέλουμε να τους καταπολεμήσουμε στους τρομοκράτες θα πρέπει να δούμε τι έγινε στη Βόρεια Ιρλανδία και τι έγινε στο Τυρόλο. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά είναι απορίας άξιων να βλέπουμε την Κίνα ε, που θεωρεί ότι ε, είναι ένα ισχυρό κράτος αλλά ταυτόχρονα νιώθει τόσο αδύναμη ως κράτος ε, που δεν σέβεται και καταστέλει ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να σέβονται τις αρχές, να ασκούν την θρησκευτική τους ελευθερία. Καταστέλει τα όνειρα των πολιτών της εάν ε, δεν ε, σε, ακολουθούν ακριβώς τη γραμμή πλεύσης ε, της ηγεσία της Κίνας και την εξάγει και όλα στην καταστολή αυτή η Κίνα. Λοιπόν, είμαστε κατά και θέλω να υπενθυμίσω και το όνομα του Ιλχάμ Τόχτη που είναι ένας επιστήμονας Ουιγούρος που εδώ και καιρό είναι υποκράτης, είναι στη φυλακή επειδή άσκησε την ελευθερία έκφρασης και αυτόν πρέπει να τον θυμόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπέλντερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι τη σήμερα ημέρα είναι ανεπιθύμητοι στο Ξινγκιάνγκ, Διότι το κομματικό κράτος της Κίνας, αυτήν ακριβώς την περιοχή είναι που δοκιμάζει αυτή την εποχή το σύστημα του εποπτείας και παρακολούθησης των ανθρώπων και χρησιμοποιεί τους Ιγούρους σαν ανθρώπινα πιόνια. Οι δυτικοί ανταποκριτέ ε, όμως καταφέρνουν που και που να μεταφέρουν κάποιες εικόνες για το τι συμβαίνει στο Ξιάνκ. Και όπως κάποιος ε, γούρους είπε ότι αυτό που εκεί λένε ασφάλεια σημαίνει ανασφάλεια για του ανθρώπου, Είπε ότι φοβάται Υπάρχουν ε, εκατοντάδες μέλη οικογενειών που υποφέρουν. Και επιπλέον, οι ε, δημόσιοι υπάλληλοι της Κίνας φαίνεται ότι είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν ε, σε φιλικές εντό αγωγικών επισκέψεις σε Ιγούρους και καταλήγουν να μένουν εκεί για καιρό και να τους παρακολουθούν. Με αυτήν λοιπόν την άγρια τη θρησκευτική της πολιτική αφομοίωσης η Κίνα οδηγεί σε παραβιάσεις. Είναι απαράδεκτο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράο τώρα έχει το λόγο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έχουν επανέλθει. Δεν μπορεί αλλιώ να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στη Σιν Γιάνγκ. Ε, αυτή η εκστρατεία στόχο έχει να εκριζώσει υποτίθεται τις τρομοκρατικές απειλές αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τις αυθαίρετες ε, κατα... Ε, φυλακίσεις στα στρατόπεδα αυτά άνθρωποι που βασανίζονται, συλλογικά τιμωρούνται και φυσικά χωρίς σωστές διαδικασίες, χωρίς δίκες αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαπράξει το <clears throat> έγκλημα να μην είναι Κινέζοι χαν. Ε, πρόκειται για μαζικές δολοφονίες, μαζικές εκτελέσεις, πρόκειται για πολύ χοντρικές ε, ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κανείς δεν επιβάλλει όρια με βάση τις αποδείξεις που υπάρχουν για τις παραβιάσεις λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σιν Γιάνγκ να καταγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση με στοχοθετημένες κυρώσεις κατά του ε, γραμματέα του κόμματος δεν μπορούν πλέον να καθυστερήσουν. κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξωτήμοι συνάδελφοι. κοινά Κίνα τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες ε, έχει αναπτυχθεί οικονομικά με εκπληκτικό τρόπο. Όμως η πρόοδος αυτή η οικονομική δυστυχώς δεν συνοδεύεται με μια αντίστοιχη πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών. Αντίθετα, αυτό που διαπιστώνουμε εδώ είναι τεράστια βήματα προς τα πίσω. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ασχοληθεί τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, έχει συντάξει και ψηφίσματα. Σήμερα, επτά ομάδες έχουν καταθέσει ένα ψήφισμα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή Σινγιάνγκ. Αυτά που ακούμε εκεί πραγματικά σχεδόν απίστευτα είναι ότι ένα εκατομμύριο σχεδόν άνθρωποι βρίσκονται σε λεγόμενα στρατόπεδα επανεκπαίδευση ε, και χρησιμοποιούνται σύγχρονα τα συστήματα τεχνολογία ε, και ουσιαστικά ε, παρακολουθούνται και οι Ουιγούροι που ζουν στο εξωτερικό. Εμεί ζητούμε από του Κινέζου να σταματήσουν τι πρακτικέ αυτέ. Δεν μπορούν να αναφέρουν το πρόσμα τη ασφάλεια, τρομοκρατία, τι αποσχιστικέ τάσει. Φυσικά υπάρχουν αυτά και κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να εγγυηθεί την εσωτερική νόμη τάξη. Όχι όμως με μέτρα που στρέφονται μαζικά κατά συγκεκριμένων θεωρητικών μειονοτήτων. Χάνει η Κίνα ε, και χάνει και σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Η Γερμανία, η βλέπουμε ότι ε, δεν ε, απελάβουν πλέον Ουγγούρου και καζάκου, διότι έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα και ζητούμε αντίστοιχα να πράξουν και τα άλλα κράτη. Εμείς υποστηρίζουμε ότι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκπροσωπούμαστε στην Κίνα σε επισκέψη εκεί να αναφέρουμε τη παραβιάση των δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να είμαστε συντηρητικοί και άτολμοι. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό το ψήφισμα και ελπίζω να αντιδράσει ανάλογα η κινησική πλευρά. Κύριε Κιούτσουκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι, λυπηρό είναι το γεγονό ότι οι μουσουλμανικέ εθνικέ μειονότητε, οι Ουγγούροι, Καζάκοι στην ε, Κίνα βασανίζονται, καταστέλνουν τα δικαιώματά του, μπορούν να ασχίσουν στη του ελευθερία. Δεν μπορεί κανεί να δικαιολογήσει τι αυθαίρετε κρατήσει ή τι εξαφανίσει ενό εκατομμυρίου ανθρώπων που είναι αθώοι άνθρωποι, αδερφοί, αδερφέ, ε, πατέρες, μητέρες που έχουν εξαφανιστεί από τις οικογένειές τους. Ε, τι γίνεται στα στρατόπεδα πανεκπαίδευση αυτά. Ε, τα παιδιά από ό,τι φαίνεται τα χωρίζουν από τις οικογένειές τους. Ε, δεν μπορούμε εμείς να, σιωπηλούμε, να σιωπούμε συγγνώμη, απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Ζητώ άμεση απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται ε, αυθαίρετα σε στρατόπεδα εγκλισμού και για την απελευθέρωση των κρατουμένων όπως ο Ιλχάμ Τόχτη, ε, που είναι πολιτικοί κρατούμενη. Ζητούμε συγκεκριμένη δράση, ζητούμε απαντήσεις, ανεξάρτητη έρευνα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα που βασίζεται ε, σε στοιχεία ε, ε, τόσο αμερικά, όπως η Εκτελεστική Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου, οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κύριες δυνάμεις τους να συγκρουστούν με χώρες που, που διεκδικούν τη δική τους κυριαρχία. Πρόκειται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η παρέμβαση τέτοιου είδους. Είναι μια υποκριτική κατάσταση. Κάνουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ διαχειριζόμαστε ε, πολέμους και παρεμβαίνουμε σε πολέμους, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, τροφοδοτώντας τους τρομοκράτες που σοβούν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εδώ το Κοινοβούλιο δεν έχουν ε, το θεμητό ε, ρόλο να μιλήσουν για ανθρώπινα δικαιώματα, για το κοινωνικό πρόγραμμα της Κίνας και για το δικό τους ρόλο, τον πολιτικό και τον οικονομικό, που είναι ο βασικός, ε, ε, τη μετατρέπουν σε βασικό ε, αντίπαλο του υπεριαλισμού. Αυτή είναι η συζήτηση η σημερινή. Ευχαριστούμε πολύ. Να μιλάτε πιο αργά παρακαλώ για να μπορούν να σας παρακολουθήσουν διερμηνείς. Ο κύριος Στόκης τώρα δύο λεπτά. Εισαγωγικά θέλω να χαιρετήσω εδώ τα θεωρία τον κύριο Ντολκονίσα που είναι ο πρόεδρος του Γουριανού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ουιγούρων. Καλώς ήρθατε. Κύριε Κούλεγαρ. Πρέπει να πω ότι το Σεπτέμβριο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε το ΕΛΚ την έκθεση για τις σχέσεις με την Κίνα. Και το έγγραφο αυτό υπογραμμίζει την στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, ότι βασίζεται σε αρχές όπως είναι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και λέει επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η κατανόηση μεταξύ των δύο τέρων. Στο πνεύμα λοιπόν αυτού του εγγράφου υψώνω τη φωνή μου για να μιλήσω για την ε, δίωξη και την σύλληψη πάνω από ενό εκατομμυρίου Ουιγούρων. Το κομμουνιστικό κράτος της Κίνας κοινικά αρνείται ότι υπάρχουν αυτά τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι Ουιγούροι που είναι κάπου 10 εκατομμύρια, ένα ολόκληρο έθνος, ο καθένας τους βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Κάτι το οποίο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θρησκευτικά δικαιώματα κλπ. Κάτι το οποίο όμως εγγράφεται στο Κινέζικο Σύνταγμα. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν τέτοιες πολιτικές παρακολούθησης κάθε Ουιγούρου και προσπάθεια αφαίρεσης της ταυτότητάς τους. Αμοιβαία εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρχει και μπορούμε να μιλάμε για αυτήν μόνον εφόσον η Κίνα διασφαλίσει σε κάθε πολίτη και ε, σε αυτούς που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες εφόσον τους εξασφαλίσει λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Θα είμαστε κι εμείς κατά της Κίνας αυτό. Οι οικονομικά συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την εταιρική αυτή σχέση δεν μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε έναν ειλικρινή διάλογο και στη... να ξεχάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε, κύριο Σκέλαν, εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Κίνα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τις μειονότητες της γιατί είναι το μεγαλύτερο έθνο στον κόσμο. Οπότε δεν βλέπω γιατί μόνο 11 εκατομμύρια που είναι οι Γούροι είναι θύματα συνεχών διώξεων και καταπίεσης. Τους ε, ενοχλούν στην πολιτιστική τους έκφραση, την ταυτότητά τους κτλ. Γίνεται πλήση κεφάλων. Λοιπόν, ζητάμε από την κυβέρνηση του Πεκίνου να σταματήσει τέτοιες πρακτικές αυθαίρετων συλλήψεων σε βάρος των μελών της μειονότητας των Ιγούρων. Ζητούμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να παρακολουθήσουν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να το θέτουν κάθε φορά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ζητούμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πιέσουν την Κίνα να σταματήσει τις παρενοχλήσεις και να μην επιτρέψουν η Κίνα να πιέζει τους Ιγούρους που βρίσκονται εκτός Κίνας να επιστρέψουν στην Κίνα. Ευχαριστούμε εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα. Τζουφρίντα. Δυστυχώς μιλάμε για επανειλημμένα περιστατικά τα οποία καταγγέλουν όχι μόνο διεθνούς φήμε δημοσιογράφοι αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συχνά και εμείς καταγγέλουμε πολύ βαριές, καταγγέλουμε πολύ βαριές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κάτοικοι του Ζιάνγκ υπόκεινται σε καθημερινούς αστυνομικού ε, ε, αστυνομικούς ελέγχους και αναγνώριση ε, προσώπου και μάλιστα τώρα επιβεβαιώνεται και η ύπαρξη ε, στρατοπέδων ε, ε, μαζικών. Φαίνεται πως γίνεται δε δίωξη των Ουιγούρων και αυτό γιατί η Κίνα εφαρμόζει ακόμα το θενατική ποινή και ο κανο... η μονομοθεσία πολυτρομοκρατίας το δικαιολογεί και μπορεί να αυθαίρετα να επιβάλλουν αυτή την νομοθεσία. Εμείς θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων, δηλαδή των Ουιγούρων και να καλέσουμε τις τρίτες χώρες προσεκτικά να εξετάσουν τα αιτήματα διεθνούς προστασίας όπως και για τις άλλες μειονότητες όπως αυτή στην περιοχή Καζάχ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντέμες Μάκερ τώρα. Οι σκέψεις είναι ελεύθερες. Ποιος μπορεί να τις εμποδίσει. Έτσι ξεκινάει ένα από τα πιο παλιά γερμανικά τραγουδάκια διαμαρτυρίας που μιλάει για την ελευθερία. Οι Κινέζοι ηγέτε πρέπει να το ξέρουν ότι δεν μπορεί κανείς να πιέσει τι σκέψει. Και όμως αυτό προσπαθούν να κάνουν στην περιοχή του Ξινγιάνγκ με το κυνήγι μαγισσών που κάνουν σε οτιδήποτε δεν είναι κινέζικο. Οι Ιγούροι λοιπόν, οι Καζάκοι διώκονται και κλείνονται σε αναμορφωτήρια. Και εκεί τους γίνεται πλήση κεφάλου μέχρι να θεραπευτούν εντό αγωγικών από την ιδεολογική τους ασθένεια και να καθαρίσουν πάλι εντό αγωγικών η σκέψη του. Ακόμα και εκτός των αναμορφωτηρίων υπάρχει εκφοβισμός των ανθρώπων, ε, απομονώνονται, τους κατασκοπεύουν. Η Κίνα από τη μια μεν είναι ανοιχτή στον κόσμο, έτσι παριστάνει, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα σκληρό κράτος και παρά τις διάφορες συμφωνίες, διαλόγους κλπ. βρίσκεται πολύ κάτω στον δίκτυο ανθρώπινων ελευθεριών. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να πιέσει τις κινησικές αρχές να σταματήσουν τις διώξεις, τις φυλακίσεις και τα αναμορφωτήρια να τα κλείσουν. Οι σκέψεις είναι ελεύθερες και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να τις εμποδίσει. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πάιτ τώρα εκ μέρους της Αλτή για ένα λεπτό ευχαριστώ. Τελευταία, η διεθνή κοινότητα έχει στρέψει του προσβολή μακριά από τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα για κάποιου ε, πραγματικού, ρεαλιστικού λόγου. Όμω, η Κίνα που θέλει να είναι οικονομική δύναμη δεν θα πρέπει να τη επιτρέπεται να παραβιάσει τα δικαιώματα των πολιτών τη. Με βάση τον ΟΗΕ, πάνω από ένα εκατομμύριο Ιγούροι κρατούνται ε, σε στρατόπεδα εγκλισμού, χωρίς να έχουν καμία πρόσβαση στους, ε, σε αυτούς οι συγγενείς τους. Ε, ε συλλέγονται δείγματα DNA, υπάρχουν ε, συστήματα παρακολούθησης GPS που καθίστανται και στα κινητά τους και στα αυτοκίνητά τους, κάμερες που βάζουν στα σπίτια τους. Κάποιοι είναι ουσιαστικά σαν να είναι όλοι σε κατοίκον περιορισμό. Υπάρχουν αυθαίρετες κρατήσεις σε στρατόπεδα εγκλισμών. Δεν ε, γίνεται λόγος για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική από την Κίνα. Πρέπει η Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέβαλε ε, προσχωρώντας ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΑΕΕ, προσυπογράφοντας τις συνθήκες και πρέπει να υπάρξει έντονη καταδίκη αυτό των πρακτικών. Κύριο Καστάλδο έχει τώρα το λόγο για το EFTD. Ευχαριστώ. Κανένα δεν μπορεί να πει ούτε μία λέξη. Έπρεπε να σιωπούν, σαν να ήταν μουγκοί. Ε, φοβόντουσαν να πούν κάτι λάθος. Ε, αυτά είναι τα λόγια φρίκη του Σεϊραγκούλ Σαϊκ Τουρμπάι, πρώην ε, δάσκαλο της κινέζικης προπαγάνδας στα κέντρα πανεκπαίδευσης, δηλαδή στρατόπεδα συγκέντρωσης που είναι κρυμμένα στις ορεινές περιοχές του Σινγκιάνγκ στην Κίνα, μειονότητε Ουιγούρων και Καζάχων, αλλά και άλλοι. Δεν υπάρχουν δε δημόσιες, ε, δημόσια μητρώα των φυλακισμένων, όμως αυτά τα στρατόπεδα υπάρχουν, όπως και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, που ε, στην ουσία εξαφανίζονται. Και υπάρχει και η διασπορά αυτών, να το επιβεβαιώνει και στα κράτη-μέλη μας. Επίσης, πολλοί ενοχλούνται διαρκώς από την ε, ε, κινέζικες αρχές. Ε, εμείς θα πρέπει, ε, έχουμε την ηθική υποχρέωση να πετήσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων αυτών των αντιφρονούντων από τα στρατόπεδα κράτη συγκέντρωσης. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει business as usual με την Κίνα. Σοφαζέρ τώρα. Ευρώπη των Αθηνών περιφέρεια του Σινγιάνγκ που είχα επισκεφτεί πριν από 20 χρόνια εδώ και πολύ καιρό είναι το θέατρο ενό ένοπλου αποσχεστικού κινήματος που έχει διαπράξει πολλαπλές επιθέσεις και που τροφοδοτείται από έναν άγριο Ισλαμισμό. Υπό τέτοιε συνθήκε, ποιο είναι το κράτο που δεν θα παρακολουθούσε εξτρεμιστικά τεμένοι ή εξτρεμιστέ. Αυτό κάνει και η Κίνα. Αυτοί όμως που μιλάνε για στρατόπεδα συγκέντρωση με 2 εκατομμύρια, χωρίς ε, επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το είπε ένας ε, από την Επιτροπή του ΟΙΕ ε, για την καταπολέμηση των βασανιστών και τα λοιπά το 2013 είναι γελία. Άκουσα 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο. Μα αυτό είναι ο μισός πληθυσμός του Παρισιού. Έτσι όμως γεννιούνται μύθοι για αυθαίρετες μαζικές κρατήσεις είναι μια ψευδής είδηση που πρέπει να την καταπολεμήσετε και όχι να την επικυρώνετε με το ψήφισμά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. σήμερα. Ακούμε ανησυχητικά πράγματα για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δράση των κινέζικων αρχών, ιδίω ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων. Καταδικάζω τι αυθαίρετε ε, ε, κρατήσει Ουιγούρων άλλων εθνοτικών μειονοτήτων, αλλά και τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων ε, προσωπικών αυτών των ανθρώπων. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στου Κινέζους ομολόγου σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ε, πρέπει να έχει άλλη προσέγγιση απέναντι στην Κίνα για να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης. Ζητώ άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων, των αυθαίρετα κρατουμένων η ελευθερία έκφραση, η θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα της ειρηνικής, των ειρηνικών συγκεντρώσεων πρέπει να επανεπιβεβαιωθούν και να τύχουν προστασία. Θα πρέπει να υπάρξει προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία, κράτος δικαίου, γιατί αυτά είναι στον πυρήνα της μακροαιωνής σχέσης Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει και η Κίνα να καταλάβει ότι είναι προ το συμφέρον τη να εφαρμόζει αυτέ τι αρχέ. Πρέπει να καταδικάσουμε την κατάσταση στην την περιοχή του Σινγκιάνγκ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόλτεκ είχε μια μπλε κάρτα ή όχι. Μάλλον για τον προηγούμενο μιλητή το ήθελε. Συγγνώμη που δεν το είδα τότε, δεν μπορώ τώρα να το κάνω. Περνάμε στον επόμενο μιλητή. Τρεμούσα η Μπασέλς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι για το ψήφισμα αυτό που αναφέρεται στις μαζικές συλλήψεις των Ιγούρων και των Χαζάκων στο Σινγιάγκ. Και χαιρετίζω και εγώ εδώ τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ιγούρων. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα των σχέσεών μα με την Κίνα. Καταδικάζει το ψήφισμα αυτό την δράση της σημερινής κυβέρνησης σε βάρος των Ιγούρων και των Καζάκων. Εμείς λοιπόν ζητάμε από την κινέζικη κυβέρνηση να σταματήσει την πρακτική αυτή των μαζικών και αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου κρατούνται άνθρωποι. Και μια ευρωπαϊκή αποστολή θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να πάει και να επισκεφτεί την περιοχή του Σινιάκ. Ζητάμε επίση από τη γηγενική κυβέρνηση να ελευθερώσει του διάφορους σιγούρους. Η Κίνα είναι πλούσια χώρα ε, και σε πόρους αλλά και σε εθνότητες. Και δεν θα πρέπει να τους φοβάται. Θα πρέπει να τους αναγνωρίσει και να τους σέβεται. Έτσι η Κίνα θα γίνει ακόμα πιο σπουδαία. Ελευθερώστε τους Ιγούρους, ελευθερώστε το Θιβέτ, ελευθερώστε την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πάρκερ τώρα. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Η κυρία Πάρκερ. Ευχαριστώ. Η Κίνα είναι ένα σημαντικό διεθνής παίκτης και έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία και για το παρόν και για το μέλλον. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι έχει και ευθύνες. Το σημερινό διεθνές σύστημα χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια και πρέπει να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και ευημερία σε όλους τους πολίτες στον κόσμο. Όμως κάποιες χώρες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα τόσο σημαντικό παίκτη λοιπόν να δείχνει ότι παραβιάζει τόσο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια ότι θέλουν ε, να αντιμετωπίσουν ε, όπως κι άλλοι τον Ισλαμικό εξτρεμισμό, αλλά η Κίνα το παρακάνει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει γενικευμένη δίωξη των ανθρώπων στο Σιντζιάνγκ. Η Κίνα πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το κοινό μας μέλλον. Η εφαρμογή και η τήρηση, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί μέρο αυτών των σχέσεων. Ευχαριστούμε, Σόγκορ. Ένα λεπτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι πολύ βασικό για μας, αλλά εκείνη έχει δείξει το χειρότερο εαυτό της. Και οι δυτικέ ε, δημοκρατίες σιωπούν, οπότε η Κίνα ε, συνεχίζει να καταπιέζει εθνικές μειονότητες, ε, βάλωτες περιπτώσεις, όπως καταπιέζει τους Τιβετιανούς, για παράδειγμα. Τώρα βλέπουμε τι συμβαίνει στην αυτόνομη περιοχή των Οιγούρων με προβακτικές εξελίξεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης κλπ. Αυτά θυμίζουν μαύρη τρύπα, όπου συσσωρεύονται οι άνθρωποι, μπαίνουν σε αυτά και δεν βγαίνουν ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να εκτιμήσει κανείς πόσες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Αυτό όμω που ξέρουμε είναι ότι κάθε οικογένεια στην περιοχή έχει έναν αγνούμενο. Άνα. Θέλαμε να αποδείξουμε πόσο αποτελεσματικό είναι ο διάλογο Κίνα και Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Χέτμαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η κατάσταση των Ουιγούρων και των Καζάχων στην επαρχία Σιντζιάνγκ της ε, ε, Κίνας ε, σημαίνει στην ουσία ένα είδος πολιτιστικής γενοκτονίας. Οι Ουιγούροι είναι συγκεντρωμένοι σε ε, στρατόπεδα. Τα παιδιά μεγαλώνουν μακριά από τις οικογένειάς τους μέσα στα σχολεία κατήχησης. Μεγαλώνουν στα ορφανοτραφεία. 13 εκατομμύρια παιδιά. Τα νούμερα είναι ε, εύγλωτα. Φανταστείτε τι γίνεται για να μπορέσουν ε, να ε, κατηχήσουν όλα αυτά τα παιδιά. Αυτά καταγγέλει η Human Rights Watch. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε από την Κινέζικη κυβέρνηση το κλείσιμο αυτών των στρατοπέδων ε, να απελευθερωθούν οι άνθρωποι που αδίκως έχουν φυλακιστεί, να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να γίνει εγγυημένα είσοδος διεθνών δημοσιογράφων ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο Catch the Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα Παρακαλώ μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά. Ε, μετά από τόσο ο κύριο Σαφχάουζερ αλλά και ο κύριο Λόπε από την Γκουε που νομίζει ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει και να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Κίνα. Κύριε Σαφχάουζερ και Γκούε, ίσως να πρέπει να έρθουν πιο κοντά γιατί λένε τα ίδια. Εγώ θέλω να μιλήσω υπέρ των δικαιωμάτων των Ουιγούρων και των Καζάχων, διότι πρόκειται για εθνοτική κάθαρση εθνοκάθαρση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε υπέρ αυτών των μειονοτήτων πρέπει να μιλήσουμε ε, ενώ θα ε, μέσω των εκπροσώπων μας που συζητούν για διάφορα θέματα. Ευχαριστώ. Κάνω για ένα λεπτό. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα κρατούσε ένα εκατομμύριο κόσμο σε στρατόπεδα και ανάγκαζε 14 εκατομμύρια κόσμο να ζουν σε κατάσταση καταστολής, θα φωνάζαμε. τουλάχιστον θα επιβάλαμε κυρώσει. Όμως, οι περισσότεροι αποφεύγουν να επικρίνουν το Πεκίνο ή να επιτύσσουν διαφάνεια για την κατάσταση που επικρατεί στη Σιντζιάνγκ, λόγω του ότι φοβούνται την οικονομική τα οικονομικά αντίπεινα. Το Κοινοβούλιο ε, πάντως ε, μιλούσε πιο ε, ανεξάρτητα. Εδώ απλά εκφράζουμε την ανησυχία μας. Ωστόσο θα πρέπει να καλέσουμε το Κίνα να κλείσει αυτά τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον όλων των ηθινών για τη δίωξη ε, αυτών των ανθρώπων και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του 21ου αιώνα. Πρέπει ως παγκόσμια κοινότητα να δράσουμε ώστε να αποφύγουμε την επόμενη μεγάλη παγκόσμια καταστροφή. Ευχαριστώ κύριος Αστρεβίτσιους. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροπε, οι μειονότητε Ουιγούρων και Καζάχων ε, και ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ συνεχώς. Ε, τεράστιες ε, οι παραβιώσεις των δικαιωμάτων, κρατήσεις, βασανιστήρια, κράτηση υποτίθεται για την επανεκπαίδευσή τους, ε, τη θρησκευτική και άλλη. Ε, πώς μπορεί να υπάρχουν τέτοια στρατόπεδα στον 21ο αιώνα. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Οι Ιγουροί και οι Καζάκοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα τον τρόπο ζωή τους να διαδίδουν ε, τη ε, πολιτισμό τους, ε, τα πιστεύω τους, τη θρησκεία τους, ενώ ταυτόχρονα είναι στην Κίνα. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε το κλείσιμο των στρατοπέδων και να το λέμε σε κάθε επόμενο πολιτικό διάλογο με την Κίνα. Είναι θέμα πρωταρχής σημασίας. Ευχαριστώ κύριο Φαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε. κάθε φορά που μιλάμε για την Κίνα ε, είναι για το θέμα τα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν τα προσθέσουμε όλα τα ψηφίσματα που έχουμε κάνει εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ε, για την παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων που ασκεί η Κινέζικη Δημοκρατία, εύκολα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα είναι ένας από τους πρωταθλητές στον κόσμο της καταστολής, του αυταρχισμού, πλάι-πλάι με τον ε, Ρωσία του Πούτιν και τη Βενεζουέλα του Νικολάς Μαδούρο. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται ακόμα περισσότερο να επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η, η, κινέζικη κυβέρνηση ε, είναι αντίθετη με το κράτος δικαίου και την ελευθερία έκφρασης. Ενώπιον ε, αυτής της κατάστασης και της καταστολής μειονοτήτων μουσουλμάνων, ε, μειονοτήτων Ιγούρων, Καζάχων και στρατοπέδων συγκέντρωση στην ε, Σιντζιάνγκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει ε, δραστήρια, να καταδικάσει αυτές τις πρακτικές και να πιέσει την Κινέζικη κυβέρνηση ώστε να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες και τις τιμωρητικές τις ενέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Σοϊντρόβα. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσαμε, η κατάσταση στο Σινιάνγκ είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι κρατούνται σε αναμορφωτήρια. Το Σινιάνγκ είναι η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο ολόκληρο. Και οι άνθρωποι αυτοί εκεί υποτίθεται ότι έχουν στηρίξει την τρομοκρατία. Ε, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κατάχρησης όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Την 1η Οκτωβρίου διαπιστώσαμε ότι υπήρξε βασική μετακίνηση οιγόρων σε οχήματα με θωρακισμένα ε, παράθυρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά κρατουμένων που μας θυμίζει την εποχή του Στάλιν. Και γι' αυτό στηρίζω την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ε, την ε, Κίνα να σταματήσει τις διώξεις αυτές. Επίσης, συμφωνώ ότι μπορούν να υπάρξουν ε, κυρώσεις κατά της Κίνας όσον αφορά αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω παρακαλώ να ζητήσω στους συναδέρφους να μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτούς που μπαίνουν στην αίθουσα. Οπότε όσο έρχεστε παρακαλώ προσέξτε κυρία Σουίτσα τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για το... και σας ευχαριστώ για το ψήφισμα αυτό, το οποίο εκφράζει τις ανησυχίες μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έπρεπε να αντικατοπρίζουν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Οι Ουιγούροι λοιπόν και οι Καζάχοι θα πρέπει να ελευθερωθούν. Συμφωνώ με το ψήφισμα. Κυρίως οι δημοσιογράφοι να ξέρετε ότι δεν έχουν δικαίωμα να πάνε σε αυτούς τους χώρους και να μεταφέρουν το τι βλέπουν. Είναι πολύ ανησυχητικό. Άλλες φορές κάτι κάνουμε. Όταν λέμε για την Κίνα δεν κάνουμε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν να συζητήσει αυτή την περίπτωση και να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ελπίζω το ψήφισμά μας να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς να ελευθερωθούν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος είναι η Επίτροπος, η κυρία Μπιακόφσκα. Πρέπει να προσέξουμε τι έχει να μας πει η Επίτροπος, οπότε ακούστε την παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την κατάσταση στο ΣΙΑΚ και ανησυχούμε πάρα πολύ από τις διάφορες αξιόπιστες αναφορές που έχουμε για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Συνάδελφοι, παρακαλώ σοπάστε και παρακολουθήστε τι λέει η Επίτροπος. Έχουμε επίσης και παρατηρήσεις από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρατσισμό κλπ. Όλα αυτά που ακούμε λοιπόν για την Κίνα είναι ανησυχητικά με τα αναμορφωτήρια, ε, γίνονται για τους Ιγούρους και άλλες μειονότητες. Τις ε, πιέσεις που γίνονται επίση στους Ιγούρους να επιστρέψουν στην Κίνα παρά τη θέλησή τους. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν κάνει έκκληση στην Κίνα να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής. Έχουμε επίσης αναφορές και από Ευρωπαίους πολίτες ε, προέλευσης από εκεί που μας λένε ότι τους πιέζουν να επιστρέψουν στην Κίνα ή πιέζουν τους συγγενείς τους εκεί. Επίσης, ε, έχουν, ε, έχει γίνει και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σε τέτοιους ανθρώπους στην Κίνα για να μην μπορέσουν να βγουν από τη χώρα και πιέσεις σε ανθρώπους από τις μειονότητες αυτές εκτός Κίνας να επιστρέψουν στην χώρα. Πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι και να ζητήσουμε το σεβασμό της αρχής της μη πίεσης για επιστροφή. Στον τελευταίο διάλογο, τον Ιούλιο του 2018, θίξαμε το θέμα της κατάστασης στο ΣΙΑΝΚ, την θρησκευτική ελευθερία, ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, κυρίως των Ιγούρων και των Θηβετιανών. Επαναλάβαμε την επιθυμία μας να υπάρξει μια διερευνητική αποστολή στο ΣΙΑΝΚ, πρόσβαση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ε, αναμόρφωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρετε ότι στηρίζει τον ύπατο εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ που ζητάει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της ε, χώρας αν θέλουμε να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να σεβόμαστε και τη θρησκευτική ελευθερία και επεπιθύσεων ε, μετακίνησης, ε, συνέρχεστε, όλες τις αρχές να μην υπάρχουν διακρίσεις. Αυτό πρέπει να ισχύει και στο Σινγιάνγκ, όπως παντού στη χώρα. Οι διεθνείς υποχρεώσεις της Κίνας διέπονται από τη διεθνή νομοθεσία. Πρέπει να επωφεληθούμε από διάλογο με την Κίνα, να είναι αυτός ανοιχτός και εμείς φροντίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη στην Επίτροπο για τη συμπεριφορά των συναδέλφων μου. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολο να κάνουν πολιτικέ δηλώσεις από το να συμπεριφέρονται κοσμίω. Κυρίσω τη λήξη τη συζήτηση και μπορούμε να προχωρήσουμε στι ψηφοφορίες. Συνάδελφοι, ας αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Βλέπω πως όλοι θέλετε να φύγετε για τα σπίτια σας νωρίς. Ο κύριος Βιώτη ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, Ζήτησα το λόγο για να καταγγείλω ένα πολύ άσχημο περιστατικό που έγινε σήμερα στην Ιταλία. Μία σημερινή εφημερίδα δημοσίευσε αυτό. Επανέρχεται η χολέρα στην ε, Νάπολη, την φέρνουν οι μετανάστες. Αυτό, το, αυτή η είδηση είναι τελείως λάθος και αειδιαστικός αυτός ο τίτλος. Εμείς καταπολεμούμε τα ψευδή νέα, τα fake news, αλλά πρέπει το Κοινοβούλιο να καταπολεμήσει αυτού του είδους τις εφημερίδες που, που ε, δημοσιεύουν μίσος και προωθούν το μίσος στην Ήπειρό μας. Είναι ντροπή τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Ο κύριος Σόσνιας ζήτησε το λόγο. Ja chciałem się powołać na artykuł 162 regulaminu e, w czasie... 276 του κανονισμού. Στη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα της βασιστικής ε, συμπεριφοράς του Πάσχου που μου αφαίρεσε το λόγο γιατί δεν ε, έλεγα πράγματα τα οποία ήθελε ε, και ήταν αντίθετα με το κόμμα του. Θα έπρεπε να είναι αντικειμενικός και να μην προεδρεύει αν δεν μπορεί. Ευχαριστώ, το σημειώνουμε. Ας περάσουμε τώρα, σας παρακαλώ, στις ψηφοφορίες να ψηφίσουμε για την ελευθερία των ε, μέσων στην Λευκορωσία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. We proceed to, uh... Περνάμε στην κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ιδιαίτερα το Αχμέτ, την κατάσταση του Αχμέτ Μανκούρ έχει ζητηθεί ονομαστική κλίση, οπότε άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. The Τέλος. Εγκρίνεται. Μαζικές αυθαίρετες ε, κρατήσεις ε, Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή Σιντζάνγκ της Κίνας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Κοέλιου για τις στρατηγικές ε, για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ πάλι με ονομαστική κλίση. The vote is closed. Τέλος. Εγκρίνεται. Congratulations. Σε χαρακτήρια κύριε Σιγητά. Τώρα προχωράμε στην ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Βος, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης Eurojust. Υπάρχει μια πρόταση ε, απόρριψη, ε, τροπολογία 195 υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Προσωρινή συμφωνία, ονομαστική κλίση. Παρακαλώ, ψηφίστε. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Φως. Έκθεση Κρίσμπεκ, αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Ε, και πάλι έχουμε πρόταση απόρριψης για την πρόταση της Επιτροπής. Την τροπολογία 146 Ποιοι είναι υπέρ της απόρριψης. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν η πρόταση. Η απόρριψη απορρίπτεται. Και πάμε στην προσωρινή συμφωνία. Παρακαλώ ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γκρίσπεκ. Ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κανονισμό θα άρει τα σφραγμού για την ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι θεσπίζουμε την πέμπτη ελευθερία εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, αγορά αγοράς, ε, αλλάξει τα δεδομένα για την ψηφιακή ε, αγορά. Ε, είναι ένα καλό παράδειγμα μιας αποτελεσματικής Ευρώπης και θέλω να σα ευχαριστήσω όλου για την υποστήριξή σα. Μάλιστα, ευχαριστούμε κυρία Κοράτσα Μπέλτ. Ψηφίζουμε για την προσωρινή συμφωνία με ονομαστική κλίση. Ποιοι... Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται αυτή η μεγάλη αλλαγή. Περνάμε τώρα την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνείς εταιρείε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ψηφίζουμε ε, για το ψήφισμα της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ανά παράγραφο θα πάμε. Παράγραφος 10. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ναι, ναι, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά βεβαίως. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 10. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Τρία κοτμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές, Νομίζω πως εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 19, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Ναι, εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Μάλιστα. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται Τα υπόλοιπα λοιπόν, οι υπόλοιπε προτάσει ψηφίσματο καταπαιτούν και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η κατάσταση στην Ιεμένη. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα για, από 7 πολιτικέ ομάδε και ο κύριο Τάνοκ ζήτησε το λόγο για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 3. Αν τον το μικρόφωνο τέλο πάντων, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μπει μετά την παράγραφο 3 το εξή καταδικάζει την τρομολόγηση δημιουργία βαλιστικών, μάλλον την χρήση βαλιστικών πυλάγων σε στόχων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων αμάχου ω στόχο ε, κατά και, τις, και είμαστε κατά τη χρήση ε, των απαγορευμένων ναρκών ε, κατά προσωπικού που Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω κανένα να βλέπω. Ναι, είναι πάνω από 40, άρα δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, να ψηφιστεί η προφορική αυτή τροπολογία και περνάμε στην παράγραφο 20 που την ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Το πρώτο ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Mm. The vote is closed. Πέρας. Adopted. Um, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά και αυτό για την παράγραφο 20 πάντα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 23 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται το λογική σκέψη τι λατινικό του αρχικού κειμένου δύο τα πρώτο ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και τώρα ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. κατά, εποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν όλα τα άλλα ψηφίσματα και περνάμε στην καταπολέμηση της τελωνιακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Υπηρεσμού, παράγραφος 1, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Adopted. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12 σε δύο τμήματα. Το πρώτο ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστικά ψηφίσμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. So, colleagues, now we can proceed. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Όμως, θέλω να σας ζητήσω, όσοι έχετε πηγαδάκια, παρακαλώ εκτός αιθούση. Αρχίζουμε με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, που είναι έκθεση του Κάρλος Κοέλιο. Ρόρι Πάλμερ είναι ο πρώτος στις επεξηγήσεις ψήφου. Έχετε το λόγο. Α, δεν είναι εδώ. Συνεχίζουμε. Η κυρία Μόνικα Μακοβέη τότε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για την ε, καταπολέμηση ατασταλιών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, από όπου βέβαια πολλοί έχουν να χάσουν. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, για το κείμενο αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Η ψηφιοποίηση των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων καθυστέρησε. Μόνο τον Ιούνιο οι χώρες μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές πλατφόρμες. Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν την διαφθορά, οι χώρες μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα ψηφιακά δελτία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη διόρθωση των εθνικών μητρών συμβάσεων και το να προσαρμοστούν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια με την ψηφιοποίηση, λιγότερη γραφειοκρατία, διευκολύνονται οι διαδικασίες, απλοποιούνται και δαπανάται με σωστό τρόπο το χρήμα των φορολογούμενων. Ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Περνάμε στον κύριο Ζαμπάσκη. Και αυτός επεξήγηση ψήφου. Παρακαλώ κύριε Ζαμπάσκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στήριξα την έκθεση του συναδέλφου Κοέλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ήδη το 2014 ένα αντίστοιχο πακέτο. Βέβαια, διάφορες χώρες είχαν δυσκολίες να υλοποιήσουν τις προτάσεις εκείνες με κυρώσεις και καταλήξαμε στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος κάποιων χωρών μελών. Τώρα λαμβάνονται υπόψη διαφορές μεταξύ των χωρών μελών γιατί χρειαζόμαστε πράγματι ευέλικτη εφαρμογή. Τώρα το πακέτο αυτό μας βοηθάει στον εξυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων. Στήριξα την έκθεση αυτή γιατί έτσι θα έχουμε online δημοσίευση ε, των όσων συμβαίνουν, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Έτσι, οι δημόσιες συμβάσεις θα γίνονται με καλύτερο τρόπο και θα υπάρχει και καλύτερος έλεγχος των δαπανών. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τζαμπάσκη. Επόμενος ομιλητής, κύριος Χωσέ Γνάσιο Αφαρία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να χαιρετήσω τον συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε όσον αφορά τις ε, δημόσιες ε, προμήθειες ε, χρειάζεται διαφάνεια ώστε να είναι αποτελεσματικές και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες. Σύμφωνα με την Κομισιόν, πολλές κρατικές προμήθειες κρίνουν την χαμηλότερη τιμή μόνο για να αναθέσουν κάποιο έργο χωρίς να κρίνουν την κοινωνικό αντίκτυπο ή την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να πάψει αυτή η κατάσταση πριν από τέσσερα χρόνια με τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου η Κομισιόν ε, επιτέλους υπέβαλε σχετικό σχέδιο να χρησιμοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας καθώς και η διασυνοριακή συνεργασία και η πλήρης αξιοποίηση της, ευρωπαϊκής, της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δημόσια ε, ρύθμιση ε, και συνεννόηση μεταξύ ιδιωτική και δημόσιου τομέα. Να αποφευχθούν καταστάσεις όπως υπήρξαν στην Πορτογαλία όπου ε, τέτοιες συνεργασίες οδήγησαν στην εκμετάλλευση πολλών εκατομμυρίων από το δημόσιο καρβανά. Ευχαριστώ κύριε Φαρία. Ε, θα πρέπει να θυμίσω σε όλους ότι η επεξήγηση ψήφου είναι για ένα λεπτό. Mr. Nekov. Yeah, ε, Ο Νέκοφ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι δημόσιε συμβάσει είναι πολύ σημαντικέ για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών σε όλε τι χώρε. Συμμερίζομαι την άποψη ότι χαμηλότερη τιμή τελικά είναι ε, το κριτήριο για την κατακύρωση των συμβάσεων. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί οι μικρότερες, ε, μάλλον οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ωφελούνται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει επίσης και το φαινόμενο αυτό της μειοδοσίας που οδηγεί σε τραγωδίες. Το είδαμε στη Βουλγαρία προσφάτως, όπου 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει ένα έργο για την παροχή γάλακτος και οπωροκυπευτικών στα σχολεία. Εκεί είχαμε απάτη, δεύτερη περίπτωση. Άρα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα πρέπει μέχρι τα τέλη του 2018 να εφαρμοστούν ηλεκτρονικές συμφάσεις. Και όταν υπάρχει απάτη, απατώνεις από τη Ευχαριστώ. Προέδρο ωραία. Ολοκληρώθηκε εδώ η επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Κοέλιο και περνάμε στην έκθεση ΦΟΣ, Οργανισμό Όποξη τη Συνεργασία στον τομέα τη ποινική δικαιοσύνη Γιώργη και θα ήθελα παρακαλώ την κυρία Μακοβέη να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τρομοκρατία, όλα αυτά γίνονται ο ρόλος της Eurojust είναι πολύ σημαντικός αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ε, συνεργασία μεταξύ των ποινικών αρχών ε, των κρατών μελών και να στηρίξουμε τις έρευνες Σε οποίες εμπλέκονται και τρίτες χώρες. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Κυρία Κύριο η Συνεργασία στον τομέα τη ποινική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Αξελφό για την πολύ καλή δουλειά του ως ε, οι, εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο και πιο ε, επιτευμένε μεθόδους. Ε, το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και οι φορείς απονόμησης δικαιοσύνης και με ενθαρρύνει η ενίσχυση του ρόλου της Eurojust για την αντιμετώπιση του ε, διασυνοριακού εγκλήματος, ανθρω, σωματεμπορία, ε, εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Είναι τομεί όπως μπορούν να ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη και Eurojust πληροφορίες για μεγαλύτερη προστασία. Το νέο εκτελεστικό, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο επίση θα βοηθήσει και ελπίζω να υπάρχουν τακτικές αναφορές και στα Εθνικά Κοινοβούλια όπως προβλέπετε. Αυτά ε, είναι σημαντικά, ιδίως για μας στην Ρηλανδία, τη διοικητική μου περιφέρεια, αλλά και για όλη την Ένωση. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει αυτή η πρόοδο στον τομέα τη συνεργασία τη Πολύ καλή δουλειά, κύριε Φω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κέλλη. Συνεχίζουμε και περνάμε στην ε, επόμενη έκθεση, που είναι η έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σόντζερτς έχει το λόγο. Αλλά φαίνεται δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Επόμενος. Η κυρία Μόνικα Μακοβέη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζω τον κανονισμό αυτό γιατί διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των διάφορων πτυχών που έχουν να κάνουν με τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλεια κλπ. Ο κανονισμός αυτός εξαφανίσει τους φραγμούς. Δηλαδή όταν δεν ε, υπάρχει αιτιολόγηση από τις εθνικές αρχές για που βρίσκονται τα δεδομένα. Υπάρχει μερικές φορές προστατευτισμός, ο οποίος όμως δεν έχει θέση στην ενιαία αγορά. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες παρατυπίες όσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των διασυνοριακών δεδομένων ή κάποιες καταχρηστικές πρακτικές που ισχύουν. Οπότε ο κανονισμός αυτός πιστεύω ότι αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος ώστε να ανοίξουν οι αγορές σε νέα μορφή εμπορίου και καινοτομίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Επόμενος, ο κύριος Πιετρόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίσαμε ένα έγγραφο για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ελεύθερης ροής των δεδομένο μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντω είναι ένα σημαντικό ζήτημα αν λάβουμε υπόψη μας την ψηφιοποίηση της οικονομίας. Στο κείμενο υπάρχει μια αρχή που καταστά δυνατή την επεξεργασία μη προσωπικών δεδομένων οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, αδικαιολόγητους περιορισμούς. Υπάρχει μια εξαίρεση που κατά τη γνώμη μου είναι ζωτική σημασία και αυτό είναι η δημόσια ασφάλεια. Λαμβάνεται υπόψη στο έγγραφο, ευτυχώ. Οπότε, όπω και άλλοι συνάδελφοι τη ομάδα μου, και εγώ στηρίζω το κείμενο αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Πιετρόφσκι. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Νεκόφα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στο σύγχρονο κόσμο οι νέες τεχνολογίες προχωρούν με τεράστια ταχύτητα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες κυκλοφορούν με λογικό τρόπο χωρίς να δημιουργούνται απειλές. Στηρίζω λοιπόν την ιδέα να επιτρέψουμε την μεταφορά των δεδομένων εκτός όντως αν υπάρχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας. Αυτή η ελεύθερη ροή θα επιτρέψει περισσότερες εξελίξεις στην καινοτομία και θα υπάρξουν περισσότερα δεδομένα και καινοτομία. Οι δημόσιες αρχές, οι δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφεληθούν τελικά από τους προμηθευτές γιατί θα υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες δεδομένων, άρα καλύτερη τιμολόγηση και καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Γι' αυτό και στήριξα την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νέκοφ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σον Κέλλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμμετείχα στην συζήτηση χτες το βράδυ για αυτό το θέμα και συστήνω το τόσο καλό έργο της Άννας Μαρία Κοράτσα Μπίλτ είναι ένα θετικό βήμα η ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς. Και χαίρομαι και για την εξαίρεση που υπάρχει για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Ο αναρμονισμός επίσης με το νέο κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι κάτι πολύ καλό. Πιστεύω ότι τα πλεονεκτήματα θα είναι πολλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν όσον αφορά τον ανταγωνισμό και θα είναι πιο εύκολο και για διάφορους οργανισμούς να αποθηκεύουν στις χώρες μέλη τα δεδομένα τους. Η Ιρλανδική οικονομία θα επωφεληθεί σημαντικά από τον περιορισμό που υπάρχει για τη δημόσια ασφάλεια. Οπότε υποστηρίζω την έκθεση αυτή. Είναι πολύ καλή η δουλειά που έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη και περνάμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για τη συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω του ΙΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Μία Πετροκόντουβα θα έχει το λόγο. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το βασικό πρόβλημα ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι τα εθνικά συστήματα δεν έρονται στο ύψος των περιστάσεων. Πολλές εταιρείε ε, φταίνε επίσης. Όταν όμως ε, παραμείνει θελοντικό το σύστημα, πάλι θα υπάρχει το ίδιο θέμα. Το κόστος είναι χαμηλό και η υγεία ή οι ζωές θα τίθενται σε κίνδυνο. Είναι καλό να γίνεται λόγος για την ε, εταιρική ευθύνη σε πολλά επίπεδα. Έχουμε πολλές ε, πολυεθνικές εταιρείες. Δεν μιλάμε όμω για δεσμευτικό ψήφισμα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να είμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή. Θέλω να ευχαριστήσω την πλειοψηφία των συμμναδέλφων που ψήφισαν υπέρ. αυτού του διεθνούς μέσου, εν αναμονή του οποίου εμείς ε, στη χώρα μου Έχουμε προωθεί την εκστρατεία για μια νομοθεσία στον τομέα της εταιρικής ευθύνης. Ε, ε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούμπολα Νάτερ. Και θαυμάζω και τους διερμηνείς που μπόρεσαν να σας παρακολουθήσουν ενώ τρέχατε τόσο πολύ. Αλλά καλύτερα να τρέχετε λιγότερο την επόμενη φορά. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος Λόλα Σάντσεθ Καλντεντέ, εξ ονόματος της ομάδος της δηλαδή ξανά της Γκουε. Δύο λεπτά θα έχετε εσείς, κυρία Καλτεντέη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που συνεπάγεται ένα ιστορικό βήμα. Ζητάμε κάτι κατεπήγον στο ψήφισμα αυτό και το λέμε στο δυνατόν πιο ρητά, πιο ρητά από πότε. Θέλουμε να είμαστε στο πλαίσιο των ΗΕ στην πρώτη θέση μισό Ένωση για μια ε, διεθνή συνθήκη που ε, θα επιβάλλει σεβασμό των δικαιωμάτων στι ε, πολυεθνικέ εταιρείε. Κάθε φορά που στον ΟΗΕ η αντιπροσωπεία τη Ένωση ή κάποιο κράτο δημιουργεί εμπόδια, κάθε φορά που τίθεται φραγμή στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα του θυμίζουμε ότι σήμερα 4 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα είπε και τα ξεκαθάρισε. Ε, η εταιρική ευθύνη δεν αρκεί ε, το σύστημα που υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθεί νομοθεσία, πρέπει να επιληθούν κυρώσεις δεν ε, ε, υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Και στρέφομαι και στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή οι εκπρόσωποι που έχουν εκλέξει πολύ σας ζητούν να κάνετε αυτή τη συνθήκη, αλλιώς δεν θα τηρήσετε, ε, μάλλον θα απογοητεύσετε τους πολίτες που δεν τους εκπροσωπείτε σωστά. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κάνουμε τη διαφορά και ελπίζω και η κυβέρνηση του Πέτρο Σάντσεθ στη Γενέβη να δραστηριοποιηθεί, να υψώσει τη φωνή του και να μην κρυφτεί πίσω από την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω έκανε η ε, κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματο. Ε, και θέλω να ευχαριστήσω του σοσιαλδημοκράτε που μα στήριξαν ε, ομόφωνα και αυτοί που δεν ψήφισαν έμειναν μόνοι του. Δεν θέλησαν να στηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω, ζητήσατε να σα πούν οι ψηφοφόροι σα τι πιστεύουν με συνθήκη. Ακόμα και η Αγία Έδρα, το Βατικανό το στηρίζει. Με τέσσερα χρόνια στο Κοινοβούλιο, βλέποντα πώ ψηφίζεται, μερικοί πραγματικά βλέπω. Ε, Ευτυχώ η πλειοψηφία ε, έχει κοινό νου, ε, έχει λογική και σήμερα ταχθήκαμε στο πλευρό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα θριάμπευσαν οι αδύναμοι αυτού του κόσμου. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για την Ιεμένη και πρώτα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γιουνούς Ομαχζέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπό Μπροστά στα μάτια των όσων δεν θέλουν να βλέπουν τι συμβαίνει, εκτελήσεται στην Ιεμένη η πιο μεγάλη ε, ανθρώπινη καταστροφή. Ο κόσμος πεθαίνει ε, κάτω, ε, από την αδιαφορία των δυτικών και πρωτευουσών που ασχολούνται με τα δικά τους μικροπροβλήματα και που ε, συμπράττουν με το απέσχυντο καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας ντροπή, στη ΣΥΠΑ, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο που πουλούν όπλα στο Σαουδική ε, Αραβία που σκοτώνει τα παιδιά της Ιεμένης. Ντροπή σε όλους όσους εξακολουθούν να δίνουν διδάγματα σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά συνεχίζουν να εμπορεύονται με το αίμα των αθώων. Και ελπίζω πως η έκκληση που έκανε το Ευρωκοινοβούλιο κατά της πώληση όπλων ε, στη Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα εισακουστεί από τα κράτη και ειδικά από τη Γαλλία. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Μαρζέ και τώρα θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο Ρουμπάν Κρέσπο. Για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επίγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη είναι αβάσταχτη. Τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ιεμένης, 20 εκατομμύρια κόσμος κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν τη ζωή τους από την πείνα. Δεν είναι το πρώτο ψήφισμα που εγκρίναμε στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ιεμένη, όμως η κατάσταση ξεκολουθεί η ίδια, γιατί τελικά το, τα χαρτιά είναι χαρτιά. Και η πραγματικότητα είναι ότι κάποια κρατημέλη ξεκολουθούν να πουλούν όπλα στην Σαουδική Αραβία ε, ενάντια στη κοινό ψήφισμα για τον έλεγχο εξαγωγή των όπλων που ψηφίσαμε σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτές τις χώρες που έχουν τα χέρια τους λερωμένα με αίμα, ανάμεσα σε αυτές είναι η κυβέρνηση του Ραχώη, η Ισπανία και, και η κυβέρνηση του Σάντσες. Είμαστε από τους βασικούς εξαγωγείς όπλων προς την Σαουδική Αραβία. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα σε ένα ψήφισμα και να κάνει τα αντίθετα η κυβέρνηση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει αλλαγή στο παραγωγικό μας μοντέλο, ώστε η εργασία πολλών οικογενειών να μην εξαρτάται από την οικονομία του πολέμου. Να μην είναι πια μόνο και μόνο ένα παλιό χαρτό αυτά που ψηφίζουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Ούρμπαν Κρέσπο και τώρα δίνουμε το λόγο στην συνάδελφο Σοίδροβα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί στήριξα το ψήφισμα για την Ιεμένη παρά το γεγονός ότι η αριστερά μπλοκάρισε την τροπολογία του συναδέλφου Κάνοκ που επίσης ήθελε να αναφερθεί το Ιράν και η Σαουδική Αραβία σε σχέση με την Ιεμένη. Πρόκειται για ένα ψήφισμα που καταγράφει στοιχεία για την τραγική σύγκρουση και την ανθρωπιστική καταστροφή για τον πληθυσμό της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια και που πρέπει να εντατικοποιηθεί παρά το συνεχιζόμενο πόλεμο που δεν είμαστε σε θέση να σταματήσουμε. Το ψήφισμα επίσης αναφέρει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, διότι η Εμένη είναι ε, στην Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ κυρία Σοίντροβα. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Μυροσλάβ Πιετρόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η χώρα αυτή υποφέρει από τον πόλεμο και εκεί κατοικούν και χριστιανοί. Το 2018 ο Διεθνής Δίκτυς Καταστολής που δημοσιεύεται από την Open Doors καταγράφει την Ιεμένη στην ένατη θέση. Στο ψήφισμά μας ε, έχουμε καταδικάσει τη βία στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά πολιτών και υποδομών. Στο έγγραφο που όπως συντάχθηκε δυστυχώς δεν αναφέρεται άμεσα η καταστολή οποία, στην οποία υπόκεινται και οι χριστιανοί. Είμαι της άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από όλα τα μέρη της σύγκρουσης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που, τους που απορρέουν από τη διεθνή νομοθεσία, διεθνές δίκαιο και καθιστά δυνατό, δυνατή την πρόσβαση των ε, ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πιετρόφσκι. Οπότε ε, εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Διακόπτεται μέχρι τις 3. präsidentin! Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνουμε τις εργασίες της Εδρίας Ολομέλειας. Ε, τα πρακτικά της ε, σχέσης χθεσινής συνεδρίασης είναι διαθέσιμα και τα αποτελέσματα ε, των συμβολίων, Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι δεν υπάρχουν, επομένως ε, δεκτά τα πρακτικά. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής από την κυρία Κάντεμαχ και λοιπούς. Καταρχάς έχει το λόγο ως ε, συντάκτη της προφορικής ερώτησης για τέσσερα λεπτά το λόγο κύριος Πόκτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η ε, παραγωγή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής είναι το βασικό, το δεσπόζωνο μοντέλο ε, για την προμήθεια της αγοράς με φθηνά κοτόπουλα. Το 95% ε, των ε, τέτοιων κτηνοτροφίων έχουν χιλιάδες κοτόπουλα. Έχουμε δηλαδή κτηνοτροφία μεγάλης έντασης, κάτι το οποίο σίγουρα πλήττει την υγεία των ζώων αλλά και την για του ανθρώπου. Σε δεκάδες χιλιάδες γίνεται η εκτροφή αυτών των κοτόπουλων χωρίς να βλέπουν το φως της ημέρας, χωρίς να έχουν χρόνο ε, για να ε, πραγματοποιήσουν τις φυσικές ανάγκε ή τις δραστηριότητες με αποτέλεσμα να βλέπουμε δυσπλασίε, να μην μπορούν να περπατήσουν, να αναπονούν, να έχουν ε, μεγάλο άγχος. Όλα αυτά είναι λίγα συμπτώματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τη γέννησή τους μέχρι το σφαγείο αυτά τα ζώα. Και πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που εμείς στον 21ο αιώνα και στι ανεπτυγμένε χώρε ανεχόμαστε. Τα θεωρούμε κάτι κανονικό, κάτι φυσιολογικό. Αν ήξερε η κοινή γνώμη πώ ε, ε, ζουν αυτά τα ζώα, δεν νομίζω να ήθελαν να φάνε το κρέα του ε, οι άνθρωποι. Τα τελευταία χρόνια ε, κύκλο ζωή των κοτόπουλων έχει μειωθεί 49 ημέρε και το βάρος τους έχει αυξηθεί, έχει διπλασιαστεί συγκεκριμένα. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που εκολάπτονται τα αυγά πρέπει να ανεβαίνουν μέσα σε δύο μήνες, δυόμιση κιλά τη μέρα. Πραγματικά ε, κάνουμε πειράματα με τη φύση και αυτά τα πειράματα έχουν βγει εκτός ελέγχου και αυτό πρέπει να ενδιαφέρει και να ανησυχεί και ε, τους ανθρώπους αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για την ε, καλή υγεία και μεταχείριση των ζώων Λόγω αυτών όλων των καταστάσεων χρειάζεται η χρήση αντιμικροβιακών, αντιβιωτικών. Το 75% δε των αντιβιωτικών και αντιμικροβιακών φαρμάκων στον κόσμο, σύμφωνα με στατιστικές, ε, χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία και ιδίω σε αυτές τις ε, εκμεταλλεύσεις ε, με τα χιλιάδες αυτά κοτόπουλα. Και με την κατάσταση αυτή αυξάνεται η μικροβιακή αντοχή, άρα αυξάνονται αυτά τα ανθεκτικά βακτήρια όπως το καμπυλοβακτήριο, το υλικοβακτηρίδιο, η σαλμονέλα. Αυξάνει την ανθεκτικότητά στα φάρμακα και αν ε, δεν αρχίσουν να λύνουμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα θα δημιουργήσει μεγάλο ζήτημα για την ανθρωπινή υγεία, διότι δεν έχουμε βρει κάποιο καλό υποκατάστατο αντί αυτών των αντιβιωτικών. Και αν αυτό χαθεί, θα πάμε 100 χρόνια πίσω ε, σε ό,τι αφορά την ιατρική. Επίση, η κτηνοτροφία ε, προκαλεί ρήπανση λόγω αμμονίας ε, και ίσως αυτό σε κάποιους να φαίνεται δευτερεύον πρόβλημα το σύγκριμα με τα αντιβετικά. Όμως όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Θα πρέπει να πιέσουμε για μια βιώσιμη αϊφόρ κτηνοτροφία. Έχω λοιπόν προ την Κομισιόν Επόμενη ερωτήσει, Ε, θα αναλάβει δράση για να βελτιώσει την επιβολή ε, των οδηγιών σε ό,τι αφορά τη συστηματική χρήση ε, των ε, τα εξανταζόμενων που με αναπτυχθεί μεταχείριση των σύγκρουση και εκμεταλλεύσει. Ποια μετασκοπεύει να λάβει να στηρίξει ανακτών συστημάτων παραγωγή κοτόπουλων ε, για να περιλαμβάνουν μεθόδου καλύτερη αναβάτη μεταχείριση των χαμηλότερων του πληθυσμού, γλωτισμό του περιβάλλοντο, προ σε εξωτερικού περιφερμένου χώρου και καλύτερη ποιότητα του αέρα, δεδομένου αυτά τα συστήματα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των υπομπών αμμονία και να περιορίσουν την ανάγκη διάκριτη χρήση αντιμικροβιακών και να βελτιώσουν τι συνδίκε διαβίωση των ζώων. Και τρίτη ερώτηση. Πότε πρόκειται να δημοσιεύσει η Επιτροπή την έκθεση σχετικά με τι κοινωνικο-οικονομικέ επιπτώσει του υποχρεωτικού συστήματο μα για το κρέα κοτόπουλου, που στο άρθρο 5 τη 2043. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρου ε, τη Επιτροπή περιμένουμε υπομονησία να ακούσουμε την Επίτροπο. Κυρία Μπιενκόφσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Έχω αναλάβει τα καθήκοντα του κύριου Αντρουκάητη τώρα και βρίσκομαι εδώ, αλλά να ξέρετε ότι και προσωπικά εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία των ζώων και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σα. Λοιπόν, όντω η μεγάλη παραγωγή κρέατος είναι η βιομηχανία αυτή που καλύπτει 200.000 εκτροφικές μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βέβαια συζητάμε για την προστασία των ζώων, την ευημερία τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει καλό έργο και σας ευχαριστώ γι' αυτό όσον αφορά την προστασία των ζώων. Βρισκόμαστε μπροστά. Οι 28 χώρες ε, μέλη εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κάθε μέρα. Το θέμα της προστασίας των ζώων το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και φροντίζουμε να βελτιώνουμε καθημερινά την ζωή των ζώων μέσω της νομοθεσίας μας. Βέβαια θα πρέπει να τηρείται πλήρως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οδηγία για την προστασία των ε, ζώων που πάνε για την κρεατοπαραγωγή. Η οδηγία αυτή λοιπόν προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο στις χώρες μέλη και έτσι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Βέβαια, η οδηγία αυτή ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία που βάζει δείκτες για την προστασία των ζώων προκειμένου να ελέγχουμε την κατάσταση. Οι πληροφορίες και οι έρευνες που έχουν δείχνουν ότι η χρήση των δικτών αυτών όπως ε, δερματίτιδες στα πουλερικά έχει οδηγήσει σε βελτιώσεις σε όλες τις εκτροφικές μονάδες. Και αυτό μας ενθαρρύνει. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε δείκτες για την προστασία των ζώων και να βελτιώνουμε συνεχώς τις ε, συνθήκες διαβίωσής τους. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για βελτίωση, πάντως η δουλειά που ήδη γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και πολύ περισσότερα. Το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους θα συνεργαστούν για να εντοπιστούν επιπλέον δείκτες όσον αφορά τα ζώα που πηγαίνουν για κρετοπαραγωγή. Τέτοιοι δείκτε μπορούν να είναι χρήσιμοι στι εθνικές αρχές αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στοχεύσει καλύτερα τη δράση τη και έτσι να εφαρμοστεί καλύτερα η οδηγία. Βέβαια, οι επενδύσει στην υγεία και στην ευημερία των ζώων ε, φέρνει και άλλα πλεονεκτήματα και ωφέλη. Και αναφέρθηκαν. Βελτιώνεται η κτηνοτροφία, ε, μειώνεται η χρήση φαρμάκων και αντιβιωτικών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε και την ε, μικροβιακή αντοχή. Η οδηγία δίνει κίνητρα για την ε, στήριξη της προστασίας των ζώων. Έχουμε κατάλογο όρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ε, εκτροφή πουλερικών. Πρόκειται για ελευθερία των ζώων να μπορούν να βρίσκονται στο εξωτερικό, ακόμα και σε περιφρεγμένους χώρους. Επιπλέον μπορούμε να συγχρηματοδοτήσουμε επενδύσεις σε συστήματα παραγωγής φιλικών προς, τον, προς τα ζώα. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση των χώρων στους οποίους ε, κρατούνται τα ζώα. Όσον αφορά το θέμα της υποχρεωτικής σήμανσης ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής, αυτή την εποχή έχουμε μία μελέτη και κάνουμε διαβούλευση με τους διαφερόμενους φορείς. Υπάρχει και έκθεση επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που εγκρίθηκε και λέει ότι η υποχρεωτική σήμανση εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία. Η εφαρμογή και τήρηση των προδιαγραφών συνεχίζεται. Το 2019 θα αρχίσουμε το έργο μας για κέντρα αναφοράς όσον αφορά την εκτροφή πουλωρικών και κουνελιών. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε επιστημονικές πληροφορίες ώστε να στηρίξουμε τις χώρες μέλη στην εφαρμογή των κανόνων για την ε, προστασία και ευημερία των ζώων. Προσβλέπω στη συζήτηση, τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Περνάμε στους ε, εκπροσώπους πολιτικών ομάδων. Καταρχάς εκ μέρου ε, του ΕΛΚ το λόγο έχει ο κύριος Φαρία για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγκρίναμε στις 13 ε, Σεπτεμβρίου την έκθεση της συναδέλφου Κάρεν ε, Κάντεμπαχ όσον αφορά την καταπολέμηση της αντίστασης στα ε, αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε πάλι με τη χρήση των αντιβιωτικών και την εντατική παραγωγή στην κτηνοτροφία κτηνοτροφίας. Ε, τα αντιβιωτικά δεν μπορούμε, ε, ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας που στόχο έχει την μείωση του κόστους και την μεγαλύτερη κερδοφορία. Η αλήθεια είναι ότι η εντατική παραγωγή χρησιμοποιεί τα αντιβιωτικά και άλλες ε, ουσίες ε, στην ε, μαζική παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή πτηνών. Αυτές οι συνθήκες επιδεινώνονται από γιατί ε, αποδυναμώνονται το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων. Έχουν προβλήματα ε, υγείας τα οποία αναφέρονται ε, και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και ε, στον άνθρωπο. Επίσης ε, θα πρέπει να αποφεύγονται βέβαια οι ασθένειες αλλά και το ίδιο και τα μικρόβια αλλά με πρακτικές διαχωρισμού και των ζώων και ευημερία των ζώων. Η δημόσια υγεία ε, περνά από την εκτινοτροφία υψηλή ποιότητα με ζώα που, τα οποία μεγαλώνουν φυσιολογικά. Θα πρέπει να σέβονται τις ανάγκες ε, των ε, ζώων και γιατί διαφορετικά αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης των ασθενειών μπορούν τα κράτη-μέλη να βασίζονται στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ώστε στις αγορές μας να φτάνουν ζωικά προϊόντα ποιοτικά που να μην είναι γεμάτα αντιβιωτικά. Και τέλος, μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταναλώνουν ε, κοτόπουλα βιομηχανικής παραγωγής χωρίς κίνδυνο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, Σοσιαλιστών Δημοκρατών, Κυρία Νόιχελ, έχει τώρα το λόγο για τρία λεπτά. Αξιότιμη πρόεδρε και κυρία Γκέπχαρτ, αξιότιμη επίτροπη, κυρίε και κύριοι, σήμερα συζητούμε την ε, κτηνοτροφία μαζικής κλίμακας. Αν δει κανείς ε, διαφημίσεις ε, για κρέας κοτόπουλο, δείχνει έναν άλλο τρόπο ζωής, ε, για, μιλάμε για ελαφρύ ε, κουζίνα, χωρίς πολλές θερμίδες, φαγητό, πολύ γινό φαγητό. Όμως πουθενά δεν αναφέρεται η πραγματικότητα. Ε, το ε, τελείω αντίθετο ισχύει με τι τη Αν ήξεραν αυτά τα ελαφρά, τα υγιεινά προϊόντα που και πώ παράγονται, δεν πρόκειται να τα κατανάλωναν οι άνθρωποι. Δηλαδή, η διαφήμιση ε, που προσπαθεί να πουλήσει τα, το κρέα κοτόπουλου καταναλωτέ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και γι' αυτό σα ερωτώ, θα κάνετε ό,τι μπορείτε, ό,τι έχετε στη διάθεσή σα μέσα να τα χρησιμοποιήσετε για να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά από ένα κομμάτι ε, κρέατο κοτόπουλου κοτόπουλο, καταλάβουν ε, πώς ε, παράγεται αυτό το, αυτό το προϊόν που δεν είναι κάτι που ε, είναι υπέρ της υγείας και ευζοίας ούτε των ζώων αλλά ούτε και υπέρ της ανθρώπινας υγείας. Ουσιαστικά σε τέτοια πτυνοτροφία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίζεται. Δεν θα έπρεπε να καταναλώνεται αυτό το κρέας. Μπορεί να είναι εύκολο να αγοράζει κανείς τέτοιο κρέας αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να ζουν έτσι τα ζώα χωρίς νερό, χωρίς αέρα, χωρίς φως γλώσσα, μέσα σε, μια, σε ένα θύλακα αμμονίας ουσιαστικά, σαν ένα θάλαμο αερίων θα έλεγα ε, για τα ζώα. Δεν μπορούν να ζήσουν έτσι αυτά τα ζώα, ε, ε, εύκολο δεν είναι καθόλου. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Εμεί θέλουμε διαφάνεια και ειλικρίνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν είναι ειλικρινέ που γίνεται τώρα. Χρειάζεται επισήμανση λοιπόν, κατάλληλη επισήμανση για να ξέρει ο κόσμο τι προϊόν αγοράζει. Όταν πηγαίνει ο αγοραστή σε ένα σούπερ χρειάζεται επισήμανση, χρειάζεται ειλικρίνη και σε ό,τι αφορά ε, τη μεταφορά, τη σφαγή, την επιλογή των διαφόρων φυλών ή ρατσών που χρησιμοποιούνται. Ε, γιατί και αυτό επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος. Αξιότιμη ε, Επίτροπε, έχετε ευθύνη, έχετε υπευθυνότητα και ε, επομένως πρέπει να δώσετε απαντήσεις και να αντιδράσετε. Ως Επιτροπή ελπίζω να αντιδράσετε και επιτέλους ε, να στραφείτε κατά αυτής της μαζικής κλίμακας πτυνοτροφίας. Γιατί είναι, θα έλεγα, η κόπρος το που πρέπει να την καθαρίσουμε ώστε να το πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Σωμάτου Συντηρητικών, ο κύριος, η κυρία Κρούπα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι πιο εύκολο να καθίσει κανείς και να εκπονήσει μια οδηγία από το να φροντίσει για την εφαρμογή της, για την τήρησή της. Υπάρχουν εκτροφικές μονάδες που θυμίζουν εργοστάσια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι δύσκολο να ξέρουμε κατά πόσο ε, τηρούνται οι προδιαγραφές προστασίας των ζώνη όχι. Πρώτα απ' όλα, φυσικές ε, συνθήκες για την εκτροφή έχουν αντικατασταθεί τώρα από βιομηχανικές εκτροφικές μονάδες. Έχουμε 8 επίπεδα κλοβών που έχουν σαν αποτέλεσμα η κτηνοτροφία να γίνεται όσο γίνεται πιο εντατικά. Τώρα μιλάμε για 32 τετραγωνικά. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι 8α4 έχει στη διάθεσή του το κάθε ζώο για να κινηθεί. Πώς ε, θα γίνει αυτό, δεν έχει πρόσβαση στο φυσικό φως και βέβαια αναπνέει αμμονία. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τα αντιβιωτικά στην εκτροφή των ζώων και να μειώσουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωση πουλερικών, γιατί κάνουν κακό στην ανθρώπινη υγεία, γιατί καταναλώνουμε και παρασιτοκτόνα και αντιβιωτικά τρώγοντας ε, πουλερικά και να μειωθεί και η ρήπανση που οφείλεται σε αυτές τις εκτροφικές ε, μονάδες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τη ζημιά που γίνεται στην ανθρώπινη υγεία και να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ανταδική κτηνοτροφία καταλήγουν στο νερό. Άρα η ρήπανση είναι τεράστια. δεν θα έπρεπε να καταλήγει η αμμονία στο νερό που στο τέλος θα καταλήξει σε ανθρώπινη κατανάλωση. Ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, των Πρασίνων και Ελεύθερη ε, Συμμαχία, ε, έτσι για 1,5 λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τρία επιχείρηματα για το, γιατί χρειάζεται κατεπηγόντω να λάβουμε δράση. Πρώτον, κτηνοτροφία ή μάλλον συγκεκριμένα πτηνοτροφία σε βάρος της καλή του υγείας υπάρχει υπερπληθισμό, συνοστισμό. Τα κοτόπουλα δεν μπορούν ούτε να ε, κουρνιάσουν, ούτε να ραμφίσουν, ε, ε, ούτε και να κινηθούν, ούτε να τεντώσουν τα φτερά τους. Αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, γίνονται εύθραυστα, ευάλωτα, με και συμπεριφορά τα ζώα. Δεύτερον, υπάρχουν επιπλοκές της υγείας και όχι μόνο για τα ζώα και για τον άνθρωπο. Υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα πτυνοτροφία εντατικής εκτροφής. Γι' αυτό την κατάσταση χρειάζεται χρήση συστηματική αντιβιωτικών για τη μείωση των συγκράτηση των επιζωτιών και των επιδημιών. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη μικροβιακή αντοχή ε, και αυτό απειλεί και τη δημόσια υγεία. Τρίτον, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις το περιβάλλον διότι η βιομηχανική εκτροφή ε, πουλερικών είναι πηγή ρήπανση. Ε, αναφέρω μία μόνο ουσία, την αμμονία που ρηπαίνει αέρα, έδαφο, ε, νερό, αντί να χρησιμοποιηθούν πρακτικέ που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο, αυτό που γίνεται είναι να χρηματοδοτούνται πρακτικέ εκμετάλλευση μακρά κλίμακα με επιδοτήσει μέσω τη κυριαρχική πολιτικής. πολιτική. Για την αντιμετώπιση των ζώων αυτή θα έπρεπε να πω το εξή. Είναι σαν ο καθρέφτη τη κοινωνία μα. Εμεί δεν θέλουμε μια κοινωνία όπου η βιομηχανική εκτροφή και η κακομεταχείριση των ζώων θα συνεχίσουν να επιδοτούνται. Μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα εκεί να κινηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, το λόγο έχει τώρα η κυρία Χάζελκαμπ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συζητάμε για την ευημερία των ζώων και των κλωσόπουλων. Ένα κοτόπουλο μεγαλώνει μέσα σε 6 εβδομάδες και από ένα κλωσόπουλο γίνεται ένα κανονικό κοτόπουλο 2 κιλών. Ε, όσο ζει με το βάρος του βουλιάζει και αυτό εμείς στην Ολλανδία αυτά το ονομάζουμε τα κοτόπουλα που εκρήγνεται. Πριν από 50 χρόνια χρειαζόντουσαν 6 μήνε τα κοτόπουλα για να ενηλικιωθούν. Τώρα σε 42 μέρε γίνεται αυτό. Σε αυτή τη σύντομη ζωή του όμω υποφέρουν. Διότι σέρνονται, έχουν διάφορα δερματικά, έχουν ακόμα και προβλήματα στην καρδιά τους. Και για να μπορέσουν να επιζήσουν όσο γίνεται περισσότερα τέτοια κοτόπουλα, γι' αυτό τους δίνουμε ένα σωρό αντιβιωτικά. Και γιατί, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει την παραγωγή και την κατανάλωση. Και αυτό σε βάρος της ανθρώπινης υγείας, σε βάρος του περιβάλλοντος και βέβαια σε βάρος των ζώων. Πρέπει να τελειώσει αυτό. Να σταματήσει αυτή η μέθοδος ταχείας ε, εκτροφής των ε, ζώων. Πρέπει να επιτρέπουμε στα ζώα αυτά να μπορούν να ζουν έξω, να βλέπουν το φως της ημέρας. Τα τελευταία 11 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοπάσει. Η έκθεσή της το δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με την ευημερία των ζώων αυτών. Αλλά δεν προτείνει καμία λύση. Βασιζόμαστε λοιπόν στους συναδέρφους και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε επιτέλους να σταματήσει αυτή η ιστορία και να προστατεύονται τα κλωσόπουλα. Έφτασε επιτέλους ο καιρός τέτοιες μέθοδοι να καταργηθούν, όπως επίσης και οι ενισχύσεις που πάνε σε τέτοιες μεθόδους εκτροφής. Ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας CFTD η κυρία Εύη. Δύο λεπτά και 30 δεύτερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, σήμερα την Παγκόσμια ημέρα των ζώων είμαι ικανοποιημένη που μπορούμε στην Ολομέλεια να συζητήσουμε αυτή την προφορική ερώτηση, κυρίως γιατί τονίζουμε εκείνα τα ζώα που πολύ συχνά τα ξεχνάμε και που αντίθετα αξίζουν την προσοχή μας. Το πρόβλημα σήμερα είναι σοβαρό και είναι σωστό το ότι το συζητάμε, διότι λένε και περισσότερες είναι οι έρευνες και οι μαρτυρίες που μας δίνουν το μέγεθος του πόσο είναι αβίωτες αυτές οι επιχειρήσεις για τη βιομηχανική παραγωγή κοτόπουλων. Ε, τα ζώα αυτά μεγαλώνουν αδύναμα με, με μόνο στόχο την παραγωγή κρέατος χαμηλής ποιότητας που πωλείται σε χαμηλές τιμές. Ε, ζουν σε φρικτές ε, καταστάσεις όπου οι ασθένειες διαδίδονται πανεύκολα. Δυστυχώς οι έρευνες που που χρησιμοποιεί η βιομηχανική παραγωγή και οι μεθόδοι που χρησιμοποιεί ε, ε, είναι ακατάλληλες ε, προληπτικά δίνουν αντιβιωτικά και αυτό δεν μπορεί να είναι μια κατάλληλη απάντηση γιατί αυτό επιδίνει, επιδεινώνει ε, το φαινόμενο της αντίστασης στα αντιβιωτικά τόσο στα πουλερικά όσο και στους ανθρώπους. Είναι πιεστικό το πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και θα ήθελα να υπογραμμίσω σε αυτό το θέμα όπως ε, θυμήσαμε το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο εκφράστηκε με την έκθεση της κυρίας Κάντεμπαχ. Γι' αυτό θεωρώ πως αυτός ο τομέας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και ότι μετατροπή των ε, κτηνοτροφικών μονάδων θα πρέπει αμέσως να γίνει σε ολόκληρη την Ένωση και στην Ιταλία πιο συγκεκριμένα που είναι η δεύτερη στη χρήση των αντιβιωτικών ε, με πάνω από 1.300 ε, τόνους αντιβιωτικών το χρόνο. Εντυπωσιακό το νούμερο. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης του κρέατος που θα βασίζεται στις σωστές πρακτικές ε, εκτροφής. Η χρήση ε, των φαρμάκων έχει μεγάλη επιρροή και στις ε, κτηνοτροφικές ομάδες. Αναφέραμε και το πρόβλημα της αμμονίας, το οποίο είναι τεράστιο και έπειτα θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και η χρήση των κλοβών. Και γι' αυτό και καλό να όλους σας να προσυπογράψετε την πρωτοβουλία των πολιτών και να ζητήσω και από την Κομισιόν να ε, νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ δηλαδή των όσων ζητούν και οι πολίτες. Ευχαριστώ εκ μέρους ε, της ομάδας ΕΝΕΦ. Μπίλτε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στριμωγμένα με τραύματα, χωρίς να μπορούν ε, να βλέπουν ε, γύρω τους, ε, χωρίς να βλέπουν καν φως της ημέρες. αυτά τα πουλερικά δεν μπορούν να ζουν υπό τέτοιες συνθήκες για να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές μας 13 δις τον παράγονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι Ιταλία μόνο το πρόβλημα. Έχουμε και στη Γαλλία ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα φαινόμενα και τα επιλέγω με τα ε, ποτόπλευτα να τα μεγαλώσουμε τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι κανονικά. Φτάνουμε στα άκρα τη γεωργική παραγωγή. Το θέμα δεν είναι να το παίζουμε vegan και ε, υγιεινολόγοι πρέπει να δούμε και άλλα θέματα. Με τη μικροβιακή αντοχή θα μπούμε σε μια πρωτάκουστη κρίση υγείας. 10 εκατομμύρια θάνατο το χρόνο το 2050. Λόγω της εντατικής χρήσης αντιμιωτικών λόγω των λοιμόξεων και των προβλημάτων ε, είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ήδη. Και έχει βέβαια και υπάρχει και το θέμα της ηθικής. Έτσι, ε, τη, ε, σε, συμπεριφερόμαστε πλέον αδύναμους. Αυτό δείχνει η κοινωνία μας ότι έχει πραγματικά ε, αποστήματα που πρέπει να σπάσουν. Δεν έχουμε άλλα μία καρδιά για τον άνθρωπο, μία καρδιά για τα ζώα, έλεγε ο Αλφόνς Δελαμαρτίν. Μία καρδιά έχουμε ή δεν έχουμε καμία καρδιά. Ακούσαμε τους ομιλητέ εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Περνάμε στου λοιπού ομιλητές με πρώτον κύριο Κέλλη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εμείς συμφωνούμε όλοι ότι το θέμα της προστασίας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και όλοι συμφωνήσαμε να μπει αυτό το θέμα στην Εμμυρίσια διάταξη. Πρέπει να δούμε τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των πουλερικών που προορίζονται σε... για ανθρώπινη κατανάλωση. Δυστυχώ όμως παρά την οδηγία που υπάρχει δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Προβλήματα είναι τα ζώα αυτά ζουν κατά δεκάδες χιλιάδες σε τραγικές συνθήκες. Δεν έχουν την ευκαιρία να συμπεριφερθούν με το φυσικό τους τρόπο, δεν έχουν την δυνατότητα για κούρνιασμα, για ράμφισμα των υποστρωμάτων εμπλουτισμού ή για να απολαύσουν το φυσικό φως. Είναι απαράδεκτο να εκτρέφουμε ζώο με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι καλό ούτε για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε πια να γνώμε. Επιπλέον, η ρήπανση εξαιτία τη βιομηχανική εκτροφή αυξάνεται και η ρήπανση από αμμονία οφείλεται ακριβώς σε αυτή την εκτροφή. Κάποια βήματα γίνονται από τον κλάδο, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να υπάρξει συνειδητοποίηση σε όλες τις χώρες για την έκταση του προβλήματος. Στηρίζω λοιπόν την Καρίν Κακέμπαχ και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει το θέμα της προστασίας των πουλερικών. Σκοπεύει να κάνει κάτι για να λυθεί το πρόβλημα. Πώς θα υπάρξει σεβασμός της οδηγίας και τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή των ζώων αυτών, αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει εκτροφή τους με αυτόν τον τρόπο στις ε, ζωές των ανθρώπων. Νομίζω ότι αν διαπιστώναμε κάτι τέτοιο για τα σκυλάκια και για τα γατάκια, θα τα είχαμε κλείσει αμέσω. Ε, Αυτέ τι μονάδε θα τι είχαμε κλείσει αμέσω. Γιατί δεν το κάνουμε και για τα πουλερικά. Σα ευχαριστώ, κύριε Βάιτ. μισή λεπτό. Σα ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, δεν ξέρω ποιος σας έγραψε την ομιλία, αλλά στην αρχή είπατε ότι η Ευρώπη ε, είναι ένας παγκόσμιος εξαγωγέας ε, πρωταγωνιστής στο τομέα της αγοράς πολυερικών. Όταν έχουμε γενετικό τροποποιημένη όχι από τη Βραζιλία που ταΐζονται αυτά τα κοτόπουλα, να μιλάμε για ευρωπαϊκή παραγωγή και θέλετε να τη διατηρήσετε για να δώσουμε στην παγκόσμια αγορά ε, τέτοια προϊόντα κρέατος όταν έχουμε ρήπανση από την αμμονία, είναι αυτό ένα μοντέλο κτηνοτροφία και κτηνοτροφία συγκεκριμένα. Μίλησατε και για θέσει εργασία. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν χιλιάδε επιχειρήσει που βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο, διότι λόγω τη διαμόρφωση των τιμών από τι μεγάλε επιχειρήσει δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν θεωρείτε ότι θα υπήρχαν περισσότερε θέσει εργασία αν άλλαζε το σύστημα αυτό το γεωργικό, αν το καταργούσαμε αυτό το ισχύον σύστημα και στηρίζαμε τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει και τι ε, ε, τους κτηνοτρόφους ε, για να προωθήσουν μια υφόρο ε, κτηνοτροφία. Βιώσιμη. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το θέλετε αυτό. Ε, δεν ξέρω. Κάποιοι που δεν ενδιαφέρονται ε, ω ζωόφιλοι για το πόσο καλά ε, με συμπεριφερόμαστε τα ζώα, α ενδιαφερθούμε για του 25.000 νεκρού που έχουμε κάθε χρόνο λόγω τη ε, μικροβιακή αντοχή. Α σκεφτούμε τον άνθρωπο. Τι άλλα επιχειρήματα θέλετε για να αλλάξετε πολιτική. και παρακαλώ, μεταπίστε και τον Επίτροπο Χόγκαν, τον αρμόδιο για τη Γεωργία, για να σταματήσει σταματήσει αυτή η βιομηχανική εκτροφή και να σταματήσει να ισχύει αυτό το μοντέλο γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Εκ, έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ε, έχουμε αυτή την εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγή όπου χρησιμοποιείται όλο και περισσότερα αντιβιωτικά. Το ίδιο θα ισχύσει και στο μέλλον γιατί χρειάζεται να γίνεται αυτό λόγω τη κακομεταχείριση ε, των ζωών που ε, γίνεται για να μπορούμε να έχουμε στο περισσότερο κρέας. Είναι τόσο χάλια οι συνθήκες διαβίωσης, εκτροφής που γι' αυτό χρειάζονται όλα αυτά τα αντιβιωτικά για να αντιμετωπιστούν οι επιδημίες, οι επιζωτίες ε, και ε, είναι μέχρι και κάποια ε, αντιβιωτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και για τον άνθρωπο. Και όλα αυτά είναι το τελευταίο που έπρεπε να γίνεται. Τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται δεν μολύνουν μόνο το κρέας των πουλερικών ε, και τα κόπρανα και τα σφάγια. Αυτό όλο, ε, το, ε, αυτά όλα πηγαίνουν έπειτα και στα ύδατα. Επομένως ρηπαίνεται το περιβάλλον, η Κομισιόν με την πολιτική που ακολουθεί, που προχωρεί με την υποστήριξη αυτών των βαρώνων στα πτυνοτροφία ουσιαστικά είναι ο υπεύθυνη για την ενίσχυση της μικροβιακής αντοχής κανείς ε, μπορούσε ε, με μια-δυο μέρες να θεραπεύσει την πνευμονία με τη χρήση αντιβιωτικών ε, και τώρα δεν γίνεται με τίποτα αυτό, διότι υπάρχουν οι νοσοκομιακές πνευμονικές λοιμώξεις, δεν βοηθάει κανένα αντιβιωτικό, δεν μπορούν να θεραπευτούν οι άνθρωποι σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ντροπή και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ βαθύ σκάνδαλο και περιμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να δραστηριωθεί γιατί αλλιώς θα πάρουμε εμείς τα χέρια μας μας ε, την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για Ζαμέ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον πρόκειται για πουλερικά για, που εκτρέφονται για κρέας, θέλω να θυμίσω, όπως το έχω επανειλημμένα ε, τονίσει στην ίντα, ότι αν ε, η χρήση τους απαγορεύεται στο 51% των κρατών μελών, παρόλα αυτά η αντιβίωση χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, ένα σωρό χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, τις οποίες πραγματεύει ο κ. Γιούγκερ και η Κομισιόν του. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται πως αυτές οι πρακτικές που χρησιμοποιούν πολύ τα φάρμακα ανταγωνίζονται και ξεπερνούν σε όγκο τις ε, συνταγές ε, που γράφονται για τους ανθρώπους. Θα πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στους όρους αυτών των εμπορικών συμφωνιών και είναι επιτακτική ανάγκη να φτιαχτεί ένα πραγματικό σύστημα ανεχνευσιμότητας και ετικετοθεσία στα εισαγόμενα προϊόντα για την ευημερία των ζώων βεβαίω, αλλά και για την ενημέρωση και τη δυνατότητα επιλογής του καταναλωτή. Γιατί και αυτό σημαίνει και ε, επηρεάζει και την υγεία των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Κύριος Ντόρφμαν, έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι εδώ συζητούμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Φαίνεται να είναι όλο και πιο αγαπητό το κρέας πουλερικό. Για τα τελευταία 10 χρόνια δούμε τα στοιχεία από 8 ε, εκατομμύρια τόνου σαν έπιασε 13 εκατομμύρια τόνου. Βέβαια, μπορούμε να συζητήσουμε για το κατά πόσον είναι θετικό αυτό. Ε, φαίνεται να καταναλώνεται περισσότερο κρέα κοτόπουλου παρά ε, μήλα, παραδείγματο χάρη στην Ευρώπη. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο αυτό είναι θετικό. Υπάρχουν ε, καταστάσει ε, και στη εκμεταλλεύσει, όπω στη Γερμανία για παράδειγμα, που προσέχουν την ευζοία των ζώων και στην Ολλανδία είχαμε επίση μια πολύ καλή συνεργασία και είδαμε και βλέπουμε και το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, πραγματικά δεν κάνει ό,τι πρέπει. Έχουμε την οδηγία 2043. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να εφαρμοστεί ε, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, μάλλον ε, θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Αν κάποιος επενδύει σε αυτά, είναι όμως πιο ακριβά τα προϊόντα του, τελικά ζημιώνεται γιατί υπάρχει ανταγωνισμός με τα άλλα. Κάποιοι έχουν εφαρμόσει σε στάβλους, σε αποθήκες ε, πιο καλά εξοπλισμένες, αλλά χάνουν γιατί υπάρχουν άλλοι οποίοι ε, φέρονται διαφορετικά και τελικά βλέπουμε, όπως και με την περίπτωση τη της παραγωγής αυγών, να παράγονται ε, στην Ουκρανία και να έρχονται δεσμολόγητα, τα αυγά για παράδειγμα ε, στην Ευρώπη. Το ίδιο γίνεται. Ε, είναι οι ίδιοι κανόνες όμως στη, με τα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν και δεν το δέχονται και οι αγρότες μας κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόρφμαν. Ήμουν λίγο πιο γενναιόδορη σήμερα με το χρόνο αγόρευσης, διότι δεν έχω πάρει καμία αίτηση για την διαδικασία Catch the Eye. Δεν ήθελα να διακόψω λοιπόν κανέναν. Και άλλωστε σχεδόν ποτέ δεν έχουμε τέτοια ομοφωνία σε όλες τις αγορεύσεις που ακούσαμε. Ε, και δεν ήθελα να τους διακόψω τους ομιλητές. Δίνω το λόγο στην Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, όσοι πήρατε το λόγο. Είναι ένα σημαντικό θέμα και σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για αυτή τη σύντομη συζήτηση θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις σας και το μήνυμά σας στον Επίτροπο Αντρουκάιτεν. Αλλά θέλω να τονίσω προηγουμένως δύο πράγματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα. Θέλει να προχωρήσει το ζήτημα και να τηρείται η οδηγία. Κατά τα άλλα και γι' αυτό οι παρατηρήσεις σας είναι πολύτιμες. Θα συνεργαστούμε για να μειωθούν οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος της βιομηχανικής εκτροφής πουλερικών. Και αυτό και υπέρ των πουλερικών, αλλά και υπέρ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Όλες τις παρατηρήσεις σας, λοιπόν, θα τις λάβουμε υπόψη. Αλλά θα σας πω και κάτι εγώ προσωπικά, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να κινητοποιήσω τα πράγματα περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Οπότε ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στο επόμενη Ολομέλεια, τη 2 του Οκτωβρίου. Τα πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη σύνοδο. Τη απουσία ενστάσεων, τα ψηφίσματα θα προωθηθούν στους αποδέκτες τους. Διακόπτεται η σύνοδος.